Good morning, everyone. I think we'll make a start. I know we weren't due to start. We're due to start, Mrs. Irigoyen Perez's. Καλημέρα σε όλους. Ε, εντάξει, έγινε, πήγε 9 και 10. Θα κάνουμε κάποιες ανακοινώσεις καταρχήν για ζέσταμα. Καλώς ορίσατε σε αυτήν την συνεδρίαση μιας ε, συνεδρίας. Ε, είμαι ευτυχής που βλέπω το μεγαλύτερο τμήμα της ομάδας μας παρών για την πρώτη έκθεση. Ο κ. Σμίτ είναι εδώ, ο κ. Ζουβάν δεν, είναι, εδώ όμως. Για να στραφώ προς το ΕΛΚ. Ναι, και τότε θα έχει έρθει και η κυρία Λίβερικ. Και, κυρία Χάνσλικ την καλωσορίζω να κάνω κάποιες ανακοινώσεις. Νομίζω ότι βγαίνουμε στο διαδίκτυο όσοι Να σας πω λοιπόν ότι στους φακέλους σας, συναδελφοί, θα βρείτε κάποιες συνοπτικές σημειώσεις για δύο από τις πρόσφατες ακροάσεις μας ε, για Έχουμε, εκεί, έχουμε εδώ την κυρία Ρέντιν και τον κύριο Ντάλι. Από ό,τι καταλάβαμε, είναι πιθανόν μέχρι το τέλη Μαΐου να έρθει η πρόταση της Κομισιόν για την ατζέντα του καταναλωτή. Δεν είναι επίσημη η ημερομηνία ακόμα, απλώς να το έχετε υπόψη Και επίσης σε μια δημόσια κοινή εκδήλωση με την Οικονομική Επιτροπή για τις οικονομικές συμβουλές που δίνουν τα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα στους καταναλωτές. Ένα πάνελ με την κυρία Μπόουρς, μια μεγάλη διάσκεψη στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επίσης για τις ωρές των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Νομίζω πως είναι θερμικό που ο ρόλος μας ως ε, ε, της προστασίας του καταναλωτή είχε αναγνωριστεί Δύο άλλα σημεία για ενημερωτικά. Μετά από την τελευταία μας συνεδρίαση, όπου ολοκληρώσαμε την ψηφοφορία για την τυποποίηση τη κυρία Κούμη, και θυμάστε ότι έγινε μια συζήτηση για το αν θα πρέπει να προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο να ζητήσουμε συμφωνία πρώτης ανάγνωσης. Η κυρία Κούμη ήρθε σε επαφή με το Συμβούλιο για να συζητήσει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και στην συνεδρία των συντονιστών στις 25 Απριλίου θα καλέσω την κυρία Κούμη να έρθει και να μας ενημερώσει, να δούμε αν συμφωνούν οι συντονιστές για να προχωρήσουμε σε αυτές τις διαπραγματεύσει και αν ναι, θα ψηφίσουμε από αυτού την επομένη στις 26 Απριλίου δηλαδή για να επιβεβαιώσουμε την εντολή. Αν συμφωνούν οι συντονιστές και το τονίζω αυτό πάντα γιατί υπάρχει μέγα ενδιαφέρον στις διαδικασίες πρώτης ανάγνωσης και εμείς ε, πολύ προσεκτικά τα παρακολουθούμε όλα αυτά με διαφανή τρόπο. Αυτά λοιπόν θα γίνουν και η κυρία Κούμη ξέρω ότι έχει έρθει το με τους κοιόδες συγητές κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Κάτι ακόμα να πω. Καταρχήν, είχαμε μια εξαιρετικά επιτυχή αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας στην Κύπρο την περασμένη εβδομάδα όπου συναντήσαμε υπουργού, συναντήσαμε τον Υπουργό Βιομηχανίας και Εμπορίου και τον Υπουργό Αρμόδιο για την Ευρώπη, για τα ευρωπαϊκά θέματα, που είναι υπεύθυνο για την γραμματεία της Προεδρίας. Έχουν φτιάξει μια γραμματεία πολύ καλή για να διευθύνει την Προεδρία και επίσης συναντήσαμε τους τέσσερις προέδρους των ειδικευμένων επιτροπών εργασίας που εργάζονται επί θεμάτων κλειδιών για τις δημόσιες προμήθειες, για την αμοιβή αναγνώριση των προσόντων, των πτυχίων, όλα τα θέματα που αφορούν τους καταναλωτές και τον, το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα αγαθά και εκείνοι μας μίλησαν μεμονωμένα. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο αυτό και επίση είχαμε μια πολύ ολοκληρωμένη παρουσίαση για τι δημόσιε προμήθειε, κρατικέ προμήθειε από μια ομάδα ειδικευμένη που εργάζεται για το, την υπηρεσία Γενικού Λογιστηρίου της Κύπρου και μας έδειξαν ένα σύστημα για ηλεκτρονικές κρατικές προμήθειες, ε, ένα top σύστημα και μας εντυπωσίασε το επίπεδο αφοσίωσης της Κυπριακής Προεδρίας. Ε, μας έδειξε πόσο σημαντικό είναι αυτές, πόσο σημαντικές είναι αυτές οι προπαρασκευαστικές επισκέψεις πριν την Προεδρία. Ήταν πραγματικά ευτυχής που μας υποδέχτηκαν πριν την Προεδρία. Και κάτι ακόμα θα ήθελα να σας πω, ότι στα τέλη του μήνα θα γίνει η διάσκεψη των Εθνικών Κοινοβουλίων, η ΚΟΖΑΚ, που οργανώνεται κοινά από τα Εθνικά Κοινοβούλια και την Διακοινοβουλευτική μας Επιτροπή και με προσκάλεσαν συγκεκριμένα να πάω και η κυρία Γκέπχαρτ θα πάει επίσης γιατί το Δανικό Κοινοβούλιο έχει ορίσει την ενιαία αγορά ως ε, θέμα κλειδί και ιδιαίτερα η εφαρμογή της οδηγίας περί υπηρεσιών. Πιστεύω λοιπόν πως η Επιτροπή μας θα είναι ευχαριστημένη και η Δανική, το Δανικό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ευχαριστήσουμε. Ε, οι συνάδελφοί μας εδώ σίγουρα θα παίξαν κάποιο ρόλο στην επιλογή της ενιαίας αγοράς ως θέματος κλειδιού για την συνάντηση αυτή και θα πάμε σύσσωμη στην Κόζακ. Τώρα, Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις που είχα να κάνω. Συγκρίνουμε επισήμω την ημερήσια διάταξη. Δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσεις. Ωραία. Και να περάσουμε. Α, ναι, να σα πω για την έγκριση των πρακτικών συνεδρία τη 28 και 29 Φεβρουαρίου. Και θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται μέχρι τα τέλη της συνεδρία εάν δεν υπάρξουν αλλαγέ. Τέλο, για το πρόγραμμα μα, ε, θα ήθελα να σα πω ότι αυτή τη στιγμή προγραμματίζουμε πρωί και απόγευμα συνεδρίαση στις 26 Απριλίου, αλλά αποφασίσαμε να ακυρώσουμε την απογευματινή συνεδρίαση λόγω του ότι αυτή τη στιγμή τα θέματα δεν είναι έτοιμα προς συζήτηση. Μόνο πρωινή συνεδρίαση 26 Απριλίου λοιπόν. 25 και 26 με συγχωρείτε, αλλά 26 θα είναι η ακρόαση για την αμοιβαία αναγνώριση προσόντων. Πολύ σημαντικό να είμαστε εδώ ε, παρόντες. Και η κυρία Βανίλη θα προεδρεύσει. Εγώ ζητώ ήδη συγγνώμη γιατί πρέπει να είμαι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά ένας από τους αντιπροέδρους θα προεδρεύσει τη συνεδρία αυτές. Υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις από συναδέλφους? Όχι, ωραία. Πολύ ωραία. Και τώρα θα εξετάσουμε τις τροπολογίες στην έκθεση της κυρίας Ιριγκουέν Πέρες. Σα δώσω το λόγο και μετά θα συζητήσουμε με του χειρότερου ηγητές. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα θα ήθελα να σας τονίσω ότι πάρα πολύ εκπλήσωμαι διότι είχαμε τόσε πρωτοπολίε στην έκθεση. Αυτό σημαίνει ότι η προστασία των καταναλωτών, των πιο ευάλωτων, είναι κάτι το οποίο δεν περνάει παρατήρητο και ότι τα μέλη τη Επιτροπή μα το ενδιαφέρον τους για το θέμα αυτό. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής για το έργο που πετέλεσαν, για τις τροπολογίες, γιατί ουσιαστικά όλες συμπληρώνουν, διευκρινίζουν την έκθεση, ξεκαθαρίζουν κάποια θέματα. Και βέβαια λόγω ε, του περιορισμένου χώρου δεν μπορέσανε όλα αυτά να τα μέσα. Πρώτα πρώτα, Έχουμε άστοχη μετάφραση και στα αγγλικά και στα γαλλικά. Ε, συμπαθάτε με, γιατί αυτό είναι κακό το να ε, έχουμε τροπολογίες ούτως ώστε να μπορέσουμε να διορθώσουμε απλώς την μετάφραση. Να σας πω τώρα για τις τροπολογίες. Θα ήθελα να αναφερθώ σε, στα εξής συγκεκριμένα θέματα. Πρώτα πρώτα, ο ορισμός του ευάλωτου καταναλωτή. Ουσιαστικά όλες οι τροπολογίες αλλιώς συμπληρώνονται. Μπορώ να τις καλύψω όλες. Η παραπομπή αυτή στην οδηγία για, τις, ε, για τους καταναλωτές, 51 και 70. Στο 70 πρόκειται για κάποια διαγραφή, ελπίζω όλοι να συμφωνήσουν και κυρίως ο κύριος Σουάμπ. Δεν είναι εδώ, τώρα εδώ. Επίσης λέμε για να υπάρξει μια στρατηγική για τους ευάλωτους καταναλωτές. Εδώ δεν μπορώ να συμφωνήσω γιατί θέλουν ε, να, να μειωθεί η προστασία των βάρων καταναλωτών. Επαναλαμβάνω. Μια τέτοια στρατηγική ποτέ θα πρέπει να οδηγήσει στο να έχουμε δύο διαφορετικά επίπεδα προστασίας ή σε περιορισμό των ατομικών ελευθεριών ή στη, στον περιορισμό των επιλογών που έχει Έχουμε την τροπολογία 78. Εδώ λέμε ότι η ρύθμιση αυτή θα χρησιμοποιηθεί από του φόρου καταναλωτέ γιατί πρόκειται για την προβλεπόμενη χρήση του ειδικού κινδύνου του φόρου καταναλωτέ και επομένω λέμε ότι όταν γίνει η τροποποίηση τη οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων να εστιαστεί στι ανωτέρω ανησυχίε. Κύριε ε, πλευρά σε λιπαρά και ζάχαρη είναι πάρα πολύ βασικό. Εδώ πέρα έχουν πάρα πολλέ ε, τροπολογίε, πρόκειται για συμπληρωματικέ. Όλοι συμπληρώνονται. Και τώρα επεξεργάζομαι μία συμβαστική τροπολογία για να καλύψει όλα αυτά τα οποία ε, προβληματίζουν τους συναδέλφους. Έχουμε την αυτορύθμιση της βιομηχανίας μια μεριά και φτάσουμε και στο ότι θα πρέπει να έχουμε μια ανάλυση για να δούμε κατά πόσον πρέπει να θεσπιστούν πιο αυστηροί κανόνες. Εν τέλει. Αύριο το απόγευμα θα λάβετε όλες τις συμβαστικές και στις 26 Απριλίου στις 10 παρατήρου θα γίνει η ψηφοφορία. Για άλλη μια φορά. Σας ευχαριστώ για την συνεργασία σας και ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε να αναβαθμίσουμε την προστασία των ευαλότερων καταναλωτών που είναι κάτι το οποίο ε, είναι θεμητό, είναι δίκαιο και να έχουμε ασφαλή, δυναμική και ανταγωνιστική αγορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος. Εμείς ευχαριστούμε. Ε, υπάρχει πρώτη προσέλευση στην συνεδριαστή μας γιατί όπως ξέρετε έχουμε και σήμερα απεργία στις δημόσιες μεταφορές. Οπότε, στο μεταξύ, ας λάβει το λόγο ο, ο, ο, ο ο, ο, συναδελφός μας, ο συγητής, ο κυριός Τελεφλής δεν είναι εδώ. Και είμαι και εγώ και ο συγητής. Thank you very much, Mr. Chairman. And, and uh, thanks to uh, the rapporteur. Smith, uh, ευχαριστώ, ευχαριστώ και την συγκέντρια. Ήδη έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα στο παρελθόν και δεν μπορώ πάνω να συμφωνήσω με τα περισσότερα από αυτά τα οποία άκουσα από την εισηγήτρια. Έχουμε επίσης την ε, έκθεση για την οποία διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις, δεν γνωρίζω δε. Εάν ε, θα δεχθεί τελικά ή όχι η εισηγήτρια όλες τις τροπολογίες για τον ορισμό Αυτό τώρα με οδηγεί στο να σας πω ότι η γενικότερη πολιτική μου άποψη δεν θα πρέπει να έχουμε υπερβολικά ευρύς ορισμού. Γιατί σε αυτή την περίπτωση όλοι θα χαρακτηριζόντουσαν ευάλωτοι καταναλωτέ. Γιατί και εγώ σε κάποιε περιπτώσει μπορώ να χαρακτηριστώ ευάλωτο. Ακόμα και ο πρόεδρό μα σε κάποιε περιπτώσει μπορεί να χαρακτηριστεί Τέτοιο καταναλωτής. Όμως δεν είναι αυτός ο στόχος της οδηγίας. Γι' αυτό σας λέω. Ας ε, είναι κάπως στενότερο ορισμός, κάπως πιο στοχευμένο. Εάν επομένω χρησιμοποιήσετε τον ε, ορισμό που αφορά το, το, το, ανήκειν σε κάποια ομάδα, ε, αυτό είναι έργο δύσκολο. Αν χρησιμοποιήσει κανεί το φίλο. Τι, όλες οι γυναίκες είναι ευάλωτες. Εδώ και πολλά χρόνια παντρεμένος. Και πολλές φορές εγώ είμαι ο ευάλωτος στο ζευγάρι. Είμαι γι' αυτό σας λέω. Νομίζω ότι είναι παρακεκινδυνευμένο όπως πανέφερα. Second, to, to claim that all consumers... Επίσης, Όλοι οι καταναλωτές, όλοι οι επιβάτες, όλοι οι πελάτες των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όλοι θα μπορούσαν να κρατήσουν ευάλωτα. Ε, αυτό είναι κίνδυνος. Από το 99 είμαι τακτικό μέλος στην Οικονομική Επιτροπή και ε, έτσι και δημιουργεί την εντύπωση ότι μπορούμε να το τους πάντες από τα πάντα. κίνδυνο. Γιατί στα χρηματοπιστωτικά, ξέρετε, Θέλουμε να προστατεύσουμε τα χρήματα των πελατών των υπηρεσιών αυτών. Τότε θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι έχουμε εξορισμό την ανασφάλεια των αποταμιεύσεων και των τοποθετήσεων, γιατί έτσι είναι εξορισμό υπάρχει εκεί πέρα ο κίνδυνο, το ρίσκο. Από την άλλη μεριά, όσο περισσότερο διγνεύει κανεί, τόσο μεγαλύτερη απόδοση. και θα έχει κανένα για τη σύνταξή του σε 25 χρόνια περισσότερα χρήματα. So um, that's actually my, my, my, my main argument. And that's... Αυτό ήταν το βασικό μου επιχείρημα. Έχω και στο πολύς και άλλων συναδέλφων σε σχέση με αυτό. Όχι, δεν ήθελα να πω ότι δεν είναι τόσο βασικό. Φυσικά και είναι είναι φυσικά, να πω σε με τις λειτουργίες της ελληνικής αγοράς, συμφωνώ με αυτό. Όμως, όπως σας είπα, έχω αυτές τις επιφυλάξεις, τις αμφιβολίες και ελπίζω ότι όταν ήρθε η ώρα των συμβιβαστικών τροπολογιών θα λάβετε υπόψη τόσο πρεσβεύω εγώ και οι άλλοι συνάδελφοι της ε, Άλντε. Εντάξει, ξέρω δεν μπορείτε να τα δεχτείτε όλα, αλλά έστω και εν μέρη. Οπότε να μπορούσαμε τελικά να τα βρούμε. Σας ευχαριστούμε, ήταν πολύ αξιόλογη και ειλικρινής η έκθεσή σας. Προερχόμαστε από διαφορετικές πολιτικές πτέρυγες του Κοινοβουλίου, ε, κάτι το οποίο βέβαια φαίνεται στη δουλειά και αυτή τη επιτροπή. Μα ήρθε και η συνάδελφος, μόλις τώρα, είσαστε έτοιμοι να το λόγο. Ναι, ναι, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ παίρνω το λόγο στη θέση του και στο όνομα του συναδέλφου Φιλίππε Ζουβά, διότι χρειάστηκε να μείνει στη Γαλλία ε, λόγω πολύ σοβαρών υποχρεώσεων. Μου διαβίβασε λοιπόν τα σχόλιά του. Θα ήθελε καταρχήν να ευχαριστήσει την κυρία εισηγήτρια, την κυρία Ερηγογέν Πέρες, που συμβάλλει στα όσα έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών. Καταρχήν, ο κ. Ζουβά θα ήθελε να υπογραμμίσει ότι υπήρξαν προβλήματα μετάφρασης στα γαλλικά του, για το σχέδιο έκθεσης και ορισμένων τροπολογιών. Ήταν ε, δύσκολη η μετάφραση. Και ενημερώθηκε και η συγγήτρια γι' αυτό επιμένει στο γεγονός ότι γνωρίζει πόσο περίπλοκο είναι το θέμα και πόσο δύσκολο είναι κανείς να το καλύψει στο σύνολό τους, κυρίως σε ένα τόσο περιορισμένο πλαίσιο όσον αφορά το χώρο που μπορεί να καταλάβει μια έκθεση πρωτοβουλία και σε αυτή την σημαντική σχέση, έκθεση μάλλον. Τώρα, επί της ουσίας, ο συνάδελφος ε, Ζουβά έχει καταθέσει κάποιες τροπολογίες που αντικατοπίζουν πέντε βασικές ανησυχίες. Πρώτον, ε, αποσαφήνιση του ορισμού του ευάλωτου καταναλωτή. να, θέλει να ξεπεράσουμε αυτόν τον ορισμό της ενδογενούς ε, αναπηρίας ή ατόμου με ειδικές ανάγκες αλλά και να λάβουμε υπόψη και την κατάσταση ε, ε, την ευάλωτη δηλαδή ε, καθορίζεται ανάμε, από μια περίπτωση προσωρινής κατάστασης που καθορίζεται από τη σχέση του ανθρώπου, του συγκεκριμένου ατόμου με το περιβάλλον του το εξωτερικό. Δηλαδή να είναι ένας ορισμός εξωγενής της, ε, του ευάλωτου χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη δηλαδή το περιβάλλον του καταναλωτή. Δεύτερον, ενίσχυση της προστασίας του ευάλωτου καταναλωτή, όπου η Ευρωπαϊκή Στρατηγική θα πρέπει να επιμείνει στη νομική προστασία του ευάλωτου καταναλωτή και άρα ενίσχυση του ίδιου του σώματος της ε, νομοθεσίας, αλλά να βασίζεται και στο θέμα, στην έννοια της χειραφέτησης του καταναλωτή, που παραπέμπει στην ικανότητα του καταναλωτή, πράγμα το οποίο συχνά συζητάμε εδώ, την ικανότητα του καταναλωτή λοιπόν να λαμβάνει αποφάσεις οι οποίες είναι σημαντικές για τον ίδιο, τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση στην ενημέρωση για τα δικαιώματά του, τη δυνατότητα να μπορεί να ιδιοποιηθεί, να καταλάβει, να εννοήσει τις πληροφορίες που λαμβάνει. Πολύ σημαντικό λέει επίσης στο ίδιο πλαίσιο η ενίσχυση των πρωτοβουλίων όπως η Ντολτσέτα, ε, δηλαδή η ενημέρωση των καταναλωτών και των επιχειρήσεων ή το δίκτυο και των κέντρων καταναλωτών, το ecc ECC-MET, το οποίο στοχεύει παντού στην, Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει τους καταναλωτές. Τρίτη Ανησυχία είναι η ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών σε σχέση με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι νέες καταχρηστικές πρακτικές που βλέπουν το φως της ημέρας όσον αφορά την ε, online, ε, την επιγραμμική διαφήμιση, την ε, διάδραση ανάμεσα στη διαφήμιση και τα κοινωνικά δίκτυα και την αντίκτυπό τους στα ευάλωτα άτομα όπως τα παιδιά. Υπάρχουν εξάλλου και όχι μόνο στα παιδιά, υπάρχουν νέες προκλήσεις με τις νέες τεχνολογίες. Τέταρτη και προτελευταία Ανησυχία είναι η προστασία των ευάλωτων καταναλωτών σε σχέση με τη συνεργασία με τις επιχειρήσεις φυσικά που πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να στηρίξουμε όλες τις πρωτοβουλίες όσον αφορά την αυτορύθμιση και τέλος αναγνώριση της αδυναμίας ύπαρξης ενός οριζόντιου ομοιόμορφου μέσου για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών λόγω της, της διαφοράς και της έλλειψης ορισμού του ευάλωτου καταναλωτή. Οπότε ο κ. Ζουβά ε, προτείνει μια προσέγγιση τομεακή, αναπερίπτωση. Πέρα από αυτές τις πέντε, που αφορούν τις πέντε κύριες ανησυχίες του, έχει καταθέσει και κάποιες τροπολογίες, όπως για παράδειγμα στην παράγραφο 16, όπου θεώρησε ότι το σχέδιο έκθεσης συνέχεια την έννοια της αγοράς και των προμηθειών με τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν ευάλωτοι καταναλωτές όπως η έλλειψη διαφάνειας τιμών ή η η σε περίπτωση αλλαγής προμηθευτή. Επίσης ήθελε να διευκρινίσει συγκεκριμενοποιήσει κάποιες προτάσεις, προτείνει να ενσωματωθεί στο η διάσταση του ευάλωτου καταναλωτή στο, στο, στο χάρτη για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για τους ευάλωτους καταναλωτές και τις ανάγκες τους και θυμίζει επίσης ένα αίτημα το οποίο έχει παλιότερα διατυπώσει σε μια έκθεση για τον αντίκτυπο της ε, διαφήμισης στον καταναλωτή Ζήτησε λοιπόν εκεί μια μελέτη για τον αντίκτυπο της ε, παραπλανητικής επιθετικής διαφήμισης στους ευάλωτους καταναλωτές, που είναι το αντικείμενο της σημερινής μας συζήτησης και ιδιαίτερα των παιδιών. Αυτά. Ε, και ολοκληρώνοντας ο κύριος Ζουβέν ε, ελπίζει πως θα μπορέσει να συμβάλλει στην εκπόνηση των συμβιβαστικών που θα βρουν σύμφωνοι την συγκήτρια και τους υπόλοιπους σκιώδεις μέχρι την ψηφοφορία για την έκθεση αυτή που νομίζω θα γίνει στα τέλη του μήνα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λίγα λόγια για τις ε, τροπολογίες μας. Ε, πρώτα απ' όλα λίγα λόγια για τους ορισμούς ευάλωτος. Ε, τι είναι ευάλωτος για να απαντήσω και στον Όλε Σμιτ. Δεν μιλάμε για κίνδυνο και ανάληψη κινδύνου, αλλά για το εάν υπάρχει πρόσβαση σε πληροφορίες, για το εάν μπορεί κανείς να αντιληφθεί τις πληροφορίες και αν μπορεί να αντιληφθεί τις συνέπειες των επιλογών του μπορεί να είναι μια κατάσταση π.χ. μια παραπλανητική συμπεριφορά την οποία μπορεί να υποστούμε όλοι ή από την κατάσταση ενός ατόμου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Να τονίσουμε πως κάποιοι είναι πιο ευάλωτοι από άλλους. Μονίμως μπορεί να πει κανείς. Όπως ανέφερε και η άνθρωποι με πνευματική αναπηρία, τα παιδιά είναι πιο ευάλωτοι. Θα θέλουμε λοιπόν να προσθέσουμε στον ευρύτατο αυτό ορισμό πως κάποιες συγκεκριμένες ομάδες είναι μονίμως ευάλωτες και πρέπει να είναι στο κέντρο της υπόθεσης αυτής. Και δεύτερον πρέπει να έχουμε μία ξεκάθαρη εικόνα του τι είναι ο ευάλωτος καταναλωτής αλλιώς δεν μπορεί να είναι χρήσιμος στους καταναλωτές στην πραγματικότητα. Οπότε από ένα φιλοσοφικό επίπεδο πρέπει να περάσουμε σε ένα πρακτικό. Δεύτερον, συμφωνούμε με τον κύριο Σωά πώς θα θέλαμε μια ανάλυση από την των παραπλανητικών και επιθετικών τακτικών, ειδικά αυτών που απευθύνονται στα παιδιά. Τρίτον, ειδικά για τον καπνό και το αλκοόλ που στοχεύει άμεσα, έμεσα τα παιδιά και τους νέους θα θέλαμε μια πανευρωπαϊκή απαγόρευση ήδη υπάρχουν χώρες που έχουν απαγόρευση για τέτοια εμπορία που απευθύνεται στους ανηλικούς νομίζω η Γαλλία <clears throat> γιατί να είναι νόμιμο εταιρείε αλκοόλ και καπνού να στοχεύουν να... τους ανήλικους τέταρτον Νομίζω πως πάλι συμφωνώ με τον κύριο Ζουβά. Θέλουμε ισχυρότερη προστασία για να αποφευχθεί η υπερβολική χρέωση στα smartphones και στο διαδίκτυο. Δεν υπάρχει καμία ρύθμιση μέχρι στιγμής, αλλά υπάρχουν πολλά παράπονα. Σας ευχαριστώ. Να δούμε αν θα τα καταφέρουμε. Uh, Thank you very much. Uh, ευχαριστώ. Άλλοι βουλευτές θέλουν να σχολιάσουν. Να πω και εγώ κάποια πράγματα γιατί είμαι και εγώ σκιώδης ε, εισηγητής από μου. Um, I agree Πρώτα απ' όλα συμφωνώ με τους ε, συναδέλφους. Πράγματι υπάρχει μια πάρα πολύ καλή βάση εδώ πέρα με τις ε, τροπολογίες. Νομίζω λοιπόν πως τώρα η κυρία Ιριγκόγεν Πέρες έχει υλικό και ο κύριος Σμιτ μας είπε πως ε, κατά περίπτωση όλοι είμαστε ε, ευάλωτοι και το θυμήθηκα αυτό στην Κύπρο την προηγούμενη εβδομάδα μου υπενθύμησαν και παραδείγματο χάρη πως ε, όσοι είναι σε διακοπές είναι επίσης ευάλωτοι σε σχέση με κάποιες υπηρεσίες παραδείγματο χάρη τη χρονομερίδια αλλά και τα νοικιαζόμενα αυτοκίνητα που ξοδεύουν πολλά λεφτά και δεν έχουν όλες τις πληροφορίες και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή προετοίμασε υλικό στα αγγλικά για τους ε, καταναλωτές και πολλά από τα παραπονά τους ήταν από ανθρώπους σε διακοπές. Οπότε συμφωνώ με αυτό το οποίο είπε η κυρία Τούρουνεν αφορά τις περιστάσεις στις οποίες βρίσκεται κάποιος και περιστάσεις μπορεί να είναι προσωρινές ή μόνιμες. Αν έχουν π.χ. χαμηλό εισόδημα, αναπηρία, αν είναι ηλικιωμένοι κτλ. Γι' αυτό δεν υπάρχει ένας γενικός ορισμός. Μιλάμε για την βελτίωση των όσων κάνουμε σε σχέση με την ομοθεσία περί καναλτών για να καλύπτει αυτά τα σημεία και χρειαζόμαστε στοχευμένη νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό ε, μπορούμε να επικεντρωθούμε στο πεδίο εφαρμογή των όσων λέει η κυρία Ριγκόγεν και να μην ε, προχωρήσουμε σε κάποιες δηλώσεις οι οποίες δεν είχαν ε, στήριξη. Ανησυχώ γιατί φεύγουμε από τα βασικά ζητήματα για την ατζέντα των καταναλωτών, γιατί υπάρχει χρόνος για αυτά ακόμα και είπαν κάποιοι συνάδελφοι πως ελπίζουν πως η ατζέντα των καταναλωτών θα ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα των ευπαθών καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν κάποια ζητήματα πρόσβασης ε, σε ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες και το τι σημαίνει αυτό σε δύο κατευθύνσεις. Ω ένα βαθμό μπορεί κάποιο να είναι ευάλωτο γιατί έχει πολλές πληροφορίες αλλά δεν ξέρει το, τι, το εάν είναι πραγματικά αμερόληπτε αυτές τι πληροφορίες και μπορεί παραδείγματο να κάνει συγκρίσει τιμών που υπάρχουν πολλά site που το κάνουν αυτό πως ξέρει κανείς ε, εάν του προσφέρεται ένα εύρο προϊόντων αυτό το συζητήσαμε χτες στην ομάδα εργασίας ψηφιακής οικονομίας της Επιτροπής μας με κάποιους λιανοπολίτες. Και νομίζω πως ένα από τα βασικά μηνύματα εδώ πέρα είναι πως πρέπει να είμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση και δεν πρόκειται για συγκεκριμένες ομάδες γιατί αλλάζουν ε, οι καταστάσεις ε, και οι περιστάσεις συνεχώς ε, ανέφερε η συνάδελφος στο παράδειγμα των κινητών τηλεφώνων. Εμείς ζητήσαμε ένα πλαφόν στους λογαριασμούς για να μην υπάρχει πρόβλημα με το roaming το οποίο εφαρμόστηκε στον πρώτο κανονισμό roaming. Τώρα ζητήσαμε το ίδιο και για τα δεδομένα. Πάλι ένα παράδειγμα όπου η έλλειψη γνώσης, η έλλειψη διαφάνειας και πληροφοριών ε, καθιστά ευάλωτους τους καταναλωτές. Επίσης ε, το ζήτημα της σύγκρισης ε, των τιμών πρέπει να μας απασχολήσει στο μέλλον. Νομίζω πως ζητήματα για την σύνδεση μεταξύ μαγαζιών στο διαδίκτυο και με φυσική παρουσία είναι σημαντικό. Ε, η διαφορά των τιμών που μπορεί να προκύψει υπήρχε η κυρία Ριγκόγιν λέει πως κάποιες τιμές είναι υψηλότερες στο ίντερνετ. Δεν νομίζω, εγώ νομίζω πως είναι χαμηλότερες. Τόσο μιλάμε και για το, εξαρτάται και από το γιατί αγαθά μιλάμε. Αλλά υπάρχουν επίσης οι δυνατότητες ε, ένας καταναλωτής να μπορέσει να παραγγείλει αγαθά μέσω του ε, ντόπιου καταστήματος ε, μέσω του διαδικτύου ε, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για όσους είναι περιορισμένοι στο σπίτι τους. Οπότε πρέπει εδώ πέρα να παράγουμε νομοθεσία που θα προστατεύει τους καταναλωτές σε όλες τις περιστάσεις μπορούμε να προβλέψουμε και στις ειδικέ περιπτώσεις. Και επανερχόμαστε βεβαίως στο όλο ζήτημα της σωστής προετοιμασίας ε, της νομοθεσίας και του να έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας ε, και παραδείγματος χάρη ναι, αυτό φάνηκε και στις εκθέσεις ε, Σβένσον και Τριανταφυλλίδη. Αυτή είναι η συνεισφορά μου που ελπίζω να είναι και ευρύτερη ε, εκ μέρους της Επιτροπής. Ε, να σας δώσω λοιπόν το λόγο για να σχολιάσετε αυτά τα οποία ακούσατε και μετά θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια. Καλημέρα και ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το εξαιρετικό της έργο και την Επιτροπή για τις πολύ καλές ε, τροπολογίες. Θα ήθελα να πω πως ε, συμφωνούμε με την ε, πολυδιάστατη αυτή πτυχή των ευπαθών ε, καταναλωτών και θα ήθελα να επιβεβαιώσω πως είναι πρόθεση να εντάξουμε την αναπηρία και όλες τις υπόλοιπες πτυχές ε, του να είναι κανείς ευάλωτος στη γενικότερη έρευνά μας γιατί γνωρίζουμε όλοι πως προσπαθούμε να βασίζομαστε σε γεγονότα και επειδή είναι σαφές πως ε, ζούμε σε μια κοινωνία που αλλάζει συνεχώς και όπως επεσήμανε και ο κύριος Χόρμπερ ε, πρέπει βεβαίως να γνωρίζουμε συνεχώς αυτές τις πτυχές πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ του τι μπορεί να αντιληφθεί ο μέσος καταναλωτής και που μπορεί να υπάρξει μια ανάγκη που θα χρειάζεται ειδικά μέτρα. Αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε. Σημείωσα επίσης πως ζητάτε μια ειδική μελέτη για την παραπλανητική διαφήμιση, ειδικά αυτή που απευθύνεται σε παιδιά και νέους. Μπορεί να το συμπεριλάβουμε σε περαιτέρω μελέτες και θα εξετάσουμε ειδικά το πώς είναι ευάλωτοι οι καταναλωτές σε συγκεκριμένες αγορές. Και εκεί είναι χρήσιμη η έκθεση γιατί επισημαίνει τομείς ε, όπου μπορεί κανείς να είναι ευάλωτος. Και συμφωνούμε με αυτά τα οποία υπόθηκαν. Χρηματοοικονομικές υπηρεσίε, μεταφορές, ενέργεια, ε, στεγαστικά δάνεια κτλ. είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε πως μπορεί και εμείς να είμαστε προσωπικά ευάλωτοι σε κάποια κατάσταση όμως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σαφείς στο ότι έχει δείξει η έρευνα πως ίσως το επίπεδο του μέσου καταναλωτή δεν ήταν αυτό το οποίο περιμέναμε ίσως ήταν Θα πρέπει λοιπόν να το δούμε αυτό στη προτινόμενα μέτρα, γι' αυτό πρέπει να συνεχίζουμε να ερευνάμε το θέμα. Και μετά θα πρέπει να δούμε πού υπάρχουν οι συγκεκριμένες ε, ευπάθειες και βεβαίως ε, θα δούμε το τι γίνεται και στα εθνικά πλαίσια, με μέτρα πληροφόρηση αλλά υπάρχει ένα όριο σε αυτά. Οπότε και η νομοθεσία είναι κάτι το οποίο πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να κάνουμε. Ε, Τέλος θα ήθελα να πω πως στους ε, τομείς που προέκυψαν ε, στην έκθεση υπάρχουν κάποια σημεία που εξετάζει η Κομισιόν το ένα είναι ο οπτικοακουστικός τομέας ε, η διαφήμιση για τα παιδιά η Κομισιόν θα επανέλθει σε αυτό θα δούμε Επίσης, το τομέα ε, της ε, ασφάλειας των προϊόντων λαμβάνεται αυτό υπόψη, αλλά μπορεί να γίνουν περισσότερα πράγματα στο σχεδιασμό των προϊόντων. Εκεί πέρα υπάρχουν ειδικοί κίνδυνοι αν μιλάμε για ασφάλεια και υγεία. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω πως συνεχίζεται η δουλειά στο τρίτο ενεργειακό πακέτο υπάρχει μια πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και θα προσπαθήσουμε να χαρτογραφήσουμε το πώς τα κράτη-μέλη ορίζουν τους ευάλωτους καταναλωτές στο τρίτο πακέτο πώς οι πρακτικές στα διάφορα κράτη-μέλη ε, έχουν αναπτυχθεί και Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό μπορεί να μιλάμε είτε για τη φτώχεια καυσίμων είτε για οτιδήποτε άλλο. Αυτό χαρτογραφούμε αυτή τη στιγμή. Στόχο έχει ε, η έκθεση να παρουσιαστεί στο φόρουμ των πολιτών για την ενέργεια αλλά αντιλαμβανόμαστε πως είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην ε, προκύψει αυτό το φθινόπωρο αλλά για το επόμενο φόρουμ γιατί είναι πολλή δουλειά το να βρούμε τις βέλτιστες ε, πρακτικές και να δούμε και τις ε, πληροφορίες. Και το τι μέτρα λαμβάνουν τα κράτη-μέλη για να προστατεύσουν τους ευάλωτους ε, καταναλωτές. Ευχαριστώ την Επιτροπή σας και εύχομαι καλή επιτυχία για την έκθεση αυτή. Και να επισημάνω πως βεβαίως οι ευάλωτοι καταναλωτές είναι μια πρόκληση που τονίζεται στη σχετική ατζέντα. Το γνωρίζει λοιπόν η Κομισιόν πως πρέπει ε, να εργαστεί από αυτού στο μέλλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα, το λόγο η κυρία Ήργογεν Πέρτ για να ολοκληρώσει το θέμα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω όλους εσάς για τα σχόλια της παρατηρήσεις σας που σίγουρα θα βελτιώσουν την έκθεση. Όπως τονίστηκε, όλοι οι συνεισηγητές τόνισαν ότι χρειάζεται να ζητηθεί ένας ορισμός του ευάλωτου καταναλωτή. Διότι έχει καταδειχθεί ότι η νομοθεσία θα πρέπει να εξελίσσεται γρηγορότερα για να προστατεύσει θα πρέπει επίση να βρούμε για και όσον αφορά τον ε, ορισμό μία συμβαστική ε, τροπολογία. Και προβληματιζόμαστε μια που όντω ο καθένα από εμά μπορεί να βρεθεί σε θέση που βάλει κάποια στιγμή στη ζωή του. Κύριε Σμιτ, τώρα, επιτρέψτε μου πρώτα πρώτα να σα συγχαρώ για την οικογένειά σα, για τη σύζυγό σα, για τον πεθερό που αναφέρατε. Επίσης, σας ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια, γιατί όντως ε, ε, είναι θετικό το ότι αναδεικνύονται οι διαφορετικές πολιτικές απόψεις και θα πρέπει πάντως να δούμε ότι όσον αφορά ε, το, το, το ευάλωτο του καταναλωτή έχουν φανεί διαφορές των επιπέδων. Ναι, ναι, ναι, ο κύριος Βέν έχει βοηθήσει πάρα πολύ, συνάδελφε, ο, μιλήσατε στη θέση του. Και όντως, μας μεταφέρατε τι ισχύει για όλες αυτές τις ε, διατάξεις του κειμένου και για την 26. Όντως θα πρέπει να έχουμε τέτοιου είδους ε, ε, νομοθεσία και να δούμε πώς θα βρούμε πάλι την χαμένη μας εμπιστοσύνη μέσω της προστασίας. Να δούμε επίσης το ότι όλοι μπορούν να καταστούμε βάλει καταναλωτέ κάποια στιγμή. Και να δούμε τι θα γίνει και με τους ανήλικους, πρόληψη, προστασία. Φυσικά και διεξάγονται και στη Γαλλία και αλλού εκστρατείε για την προστασία και στην Ισπανία. Και έχουμε τις απαγορεύσεις του καπνίσματος, ε, τις απαγορεύσεις κατανόηση αλκοολούχων κλπ. Κύριε Χάρμπορ, σας ευχαριστώ για αυτά τα οποία είπατε, γιατί όλοι μας όταν ταξιδεύουμε όντως μπορεί να αισθανθούμε, να καταστούμε ευάλωτοι και άρα χρειάζεται να πάμε προς τα εκεί όσον αφορά την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών. Και πάλι ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε κυρία Ριγκόγεν Πέρες, λέει ο Πρόεδρος. 26 Τετάρτου θα γίνει η ψηφοφορία. Μέχρι τότε είμαι σίγουρος ότι θα έχετε κατεβάσει κάποιες τροπολογίες εσείς ίδια να δούμε κατά πόσο θα μπορέσουμε να παραπέμψουμε την έκθεση στην ε, ολομέλεια του Μαΐου. Ακούσαμε και όσα μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τώρα πάμε στο επόμενο θέμα μας. Με μεγάλη μου χαρά διαπιστώνουμε ότι έχουμε παρατηρητή ή παρατηρήτρια, παρατηρητή από την Κροατία. Δεν ξέρω το ονομάζουμε το προφέρω σωστά, τέλο πάντων. Ναι, όλο ένα και περισσότερο θέλονται τώρα παρατηρήσει από τη χώρα εκείνη. Δεν ξέρω αν ε, παγίω θα έρχεστε εσεί εδώ, Πάντω, όποτε θέλετε ευχαριστώ να έρχεστε και αν θέλετε να μα ε, πείτε ε, το τι ισχύει στην Κροατία, είμαι σίγουρο ότι οι συνάδελφοι Ευχαριστώ θα σα ακούσουν. Κάνουμε τώρα μία εισήγηση Σύντομη θέλετε. Σας ευχαριστώ. Σας χαιρετώ όλους, λέει ο κύριος Μάτουσιτς. Έτσι βάζω εγώ το λιθαράκι μου στον αφορά την ευρωπαϊκή πορεία της ε, Κροατίας και επίσης έτσι να δούμε κατά πόσον ε, μπορούμε να προωθήσουμε αυτές τις ιδέες, τις προτάσεις εδώ για όλα αυτά τα θέματα το οποίο συζητάτε. Ευχαριστώ και πάλι. Πρόεδρο, Καλώ. Έχουμε κάποιο χρονικό περιθώριο γιατί ξέρω ότι θα πρέπει να οργανώσουμε την προβολή κάποιων διαφανειών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πάμε λίγο πιο νωρίς στο θέμα το επόμενο του κυρίου Κοφεράτη. αυτά τα δύο θέματα. Θα τα συζητώ δύο με τον κύριο Κοφεράτη, όμως τι να δούμε τώρα. Έχουμε και κάποια γνωμοδότηση. Αυτή η γνωμοδότηση αφορά την Επιτροπή των Μεταφορών. Και πρέπει να γνωμοδοτήσουμε επομένω όσον αφορά το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών. Χαίρομαι που θα συζητήσουμε το θέμα αυτό, διότι όπως προέκυψε χθε στην ομάδα εργασία για την ψηφιακή οικονομία. Εδώ μιλούμε για το πώ φτάνουν τα εμπορεύματα στου καταναλωτέ. Πολύ σημαντικό αυτό για την ενιαία αγορά. Και αντίστοιχα είναι σημαντικό το ότι σε συνδυασμό με την Επιτροπή Μεταφορών θα βοηθήσουμε Έχουμε τώρα από την Αρμόδια Γενική Διεύθυνση τον ε, Διευθυντή για να μας παρουσιάσει την ε, έκθεση επιπτώσεων της ε, πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όμως, κύριε Κοφράτη, θέλετε να κάνετε την εισήγηση ή θέλετε να μιλήσετε μετά την Επιτροπή. Ό,τι θέλετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω πως ίσως ήταν σκόπιμο να πω δύο λόγια στην... καταρχήν, να κάνω μια εισαγωγή και έπειτα θα δούμε και τις λεπτομέρειες. Φυσικά η συζήτηση θα αναπτυχθεί και σε επόμενες ευκαιρίες. Θα έχουμε τη δυνατότητα να εμβαθύνουμε στα διάφορα κεφάλαια. Πράγμα το οποίο δεν είναι σκόπιμο ούτε και δυνατόν σήμερα. Λοιπόν, το θέμα που μας απασχολεί, όπως λέγατε, είναι ο κανονισμός που προτείνει η Κομισιόν και που συνοψίζει τους προσανατολισμούς για την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων που πρόκειται για το σύνολο των υποδομών που μπορεί να δώσουν αν υλοποιηθούν καταλήλως σκοπεύουν, ε, σημαίνει δηλαδή αυτό αν υλοποιηθούν με την απαραίτητη ποιότητα και εγκαίρως να δώσουν στοιχεία συνοχής πάρα πολύ σημαντικά για ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης. Όπως δημήσατε και εσείς πριν από λίγο είναι πάρα πολύ σημαντικό τα αγαθά και τα άτομα να μπορούν να ταξιδεύουν όσο γίνεται πιο γρήγορα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Διότι αυτό βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσής τους και ταυτόχρονα καθιστά ανταγωνιστικά τα ε, μέρη τα οποία καλύπτονται από το δίκτυο. Η Κομισιόν έκανε μια δημόσια διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και τελικά έφτασε στην υποβολή αυτής της πρότασης που σήμερα καλούμεθα να συζητήσουμε. Εννοείται πως το δίκτυο χρειάζεται να συμπληρωθεί διότι κάποια κομμάτια ήδη έχουν αρχίσει να υλοποιούνται. Χρειάζεται να εναρμονιστεί επίσης, γιατί ανάμεσα στις διάφορες χώρες υπάρχουν ε, πολλά στοιχεία διαφορετικά και έπειτα θα πρέπει να υπάρξει μεγάλη προσοχή, να δοθεί μεγάλη προσοχή στην ποιότητα της, ε, των δομών που θέλουμε να κατασκευάσουμε αλλά και στον τρόπο κατασκευής. Θα επανέλθω σε αυτό το θέμα και γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και ελπίζω πως όλοι θα το προσέξουμε ε, δεόντως. Κατά τη γνώμη μου υπάρχει το εξής πρόβλημα. Ο εντοπισμός αυτού του δικτύου, όπως γνωρίζετε, πρόκειται για ένα διπλό δίκτυο. Δηλαδή, ένα κεντρικό δίκτυο που περιλαμβάνει τους διαδρόμους, θα πρέπει να έχουν ε, φτιαχτεί μέχρι το 2030 και έπειτα υπάρχει το γενικό δίκτυο, το ολοκληρωμένο, που θα πρέπει να έχει φτιαχτεί μέχρι το 2050. Η σημασία των διαδρόμων και η χάραξή τους έχει φτιαχτεί με βάση μια μεθοδολογία που εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να ενταχθεί στον κανονισμό για τον εξή λόγο. Δεν θα πρέπει να ε, προσπαθήσουμε να τροποποιήσουμε τα όσα ήδη έχουν καθοριστεί γιατί διαφορετικά θα καθυστερήσουμε την ε, κατασκευή του δικτύου. Όμως θα πρέπει να προσφέρουμε σε όποιον έρθει μετά από εμά τη δυνατότητα μιας μεθοδολογικής αναφοράς που θα έχει σημασία και βάρος εφόσον αποτελεί στο τμήμα του κανονισμού. Από την άποψη των υλικών επιπτώσεων, τι δεν θα άλλαζε καθόλου ο κανονισμός. Η μεθοδολογία μάλλον μέσα στον ε, κανονισμό δεν θα άλλαζε τίποτα. Νομίζω όμως ότι από πολιτικής άποψης και κυρίως ε, όσον αφορά την ομοιομορφία στο μέλλον θα ήταν κάτι το θετικό να μπει στον κανονισμό τα κριτήριο το οποίο οδήγησε στη συγκεκριμένη μεθοδολογία και στο συγκεκριμένο δίκτυο όσον αφορά την ολοκλήρωση, την εναρμόνωση, αλλά και την νέα υλοποίηση, τις νέες κατασκευές. Και νομίζω πως είναι το ίδιο σημαντικό να επιμείνουμε σε αυτό που έχει αποκληθεί η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του δικτύου. Και ως προς αυτό να τονίσω δύο, δύο υλικέ προϋποθέσεις που είναι πιο σημαντικές από τις άλλες κατά τη γνώμη μου. Η πρώτη αφορά τα διασυνοριακά τμήματα. Ένα δίκτυο που ενώνει, που συνδέει, θα πρέπει να ξεπεράσει τις υπάρχουσες διαφορές. Ε, πολύ σημαντικά σημεία είναι αυτά, εκεί όπου συναντώνται, ε, δηλαδή στα σύνορα. Έπειτα, άλλη ευκαιρία που προσφέρεται για να υπάρχουν διατροπικέ συνδέσει σε σχέση δηλαδή με την προστιθέμενη αξία. Αυτή οφείλεται στην σύνδεση μεταξύ όλων των τμήματων. Αεροδρόμια, ε, τρένα ψηλή ταχύτητα που συνδέονται με τα αεροδρόμια, τα ε, αστικά δίκτυα, σιδηρόδρομοι, αυτοκινητόδρομοι κτλ. κτλ. Κάθε κομμάτι έχει την ειδική του αξία, αλλά όταν συνδέεται με τα άλλα κομμάτια αυξάνεται η σημασία του και γι' αυτό μιλούσε για την προστιθέμενη αξία του δικτύου. Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Και έπειτα, υπάρχει κάτι ακόμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Και αυτό έχει να κάνει με το ρόλο του συντονιστή. Θα έχετε διαβάσει το κείμενο ότι για κάθε διάδρομο υποδεικνύεται και ορίζεται ένας ε, συντονιστής. Η λειτουργία του συντονιστή βασικά όπως προβλέπονται μέχρι τώρα, είναι λειτουργία επικοινωνίας, η σχέση με τους διάφορους φορείς, ε, αλλά τελικά η λειτουργία του εξαντλείται στην επικοινωνία. Δεν θέλω καθόλου να υποβαθμίσω αυτή την λειτουργία έτσι, να γίνεται η επικοινωνία όσο γίνεται πιο γρήγορα, σωστά κτλ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όμως πιστεύω πως θα πρέπει να έχουμε υψηλότερε φιλοδοξίες. Δηλαδή, ο συντονιστής να έχει την αρμοδιότητα για την επίλυση των ε, συγκρούσεων που θα μπορούσαν να προκύψουν στη διαχείριση και πριν ακόμα από την υλοποίηση του δικτύου, όταν υπάρχει μια ε, διαφορά θα πρέπει να βρεθεί ανάμεσα στα θεσμούς και στις επιχειρήσεις αλλά που θα συμμετέχουν στους φορείς δηλαδή αλλά ένας τρίτος, ένας τρίτος χωρίς να χρειάζεται δηλαδή να καταφύγουμε στην ε, πολιτική διαμεσολάβηση των κρατών αν είχαμε ένα τέτοιον συντονιστή θα έπαιζε πιστεύω πολύ σημαντικό και χρήσιμο ρόλο θα μπορούσε αυτό το ρόλο να τον παίξει ο συντονιστής ε, εμπλουτίζοντας έτσι τις λειτουργίες που ήδη του ανατίθενται με βάση το κείμενο της Επιτροπής επειδή υπάρχει ένα τελευταίο στοιχείο, όπω σα έλεγα. Υπάρχουν και άλλα σωρό άλλα προβλήματα, λεπτομερία που θα επανέλθουμε βέβαια στη συζήτηση με του συναδέλφου. Αλλά ένα τελευταίο στοιχείο που εξ αρχή ήθελα να σα αναφέρω και στην, αναφέρω και στην Επιτροπή. Όταν υλοποιούνται, κυρίω στην καινούργια κατασκευή αλλά και στην σύνδεση και στην αναδιοργάνωση. Όταν γίνονται λοιπόν μεγάλες κατασκευές, βαριές υποδομές, προκύπτει το θέμα στις σχέσεις με τις περιοχές και τους ανθρώπους. Η κατασκευή μιας σιδηροδρομικής γραμμής ή ενός αεροδρομίου γίνονται σε μέρη τα οποία είναι κατοικημένα κατοικημένες περιοχές με συνήθειες τρόπου ζωής ε, που πολλές φορές ισχύουν εδώ και αιώνε. Δεν είμαστε μπροστά σε ένα λιβάδι πράσινο όπου μπορεί να κάνει κανείς ό,τι θέλει χωρίς όμως να υπάρξουν αντιδράσεις. Παρεμβαίνουμε σε δομές πολλές φορές που είναι ήδη οργανωμένες, παγιωμένε και γι' αυτό το λόγο ο αντίκτυπος είναι επεμβατικός και συχνά ε, δημιουργεί συγκρούσεις, δυσκολίες, αντιδράσεις. Πιστεύω λοιπόν πως θα ήταν θετικό να εισαχθεί στον κανονισμό μια διαδικασία που σε κάποιες χώρες υπάρχει αλλά ε, όχι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που αφορά την αξιολόγηση των κοινωνικο-οικονομικών ε, ε, επιπτώσεων του εν λόγω έργου και έπειτα διάλογος με την περιοχή για να ε, αυληθούν οι, αυληθεί ο αντίκτυπος ώστε να μην υπάρξουν σημαντικές και μεγάλες αντιρρήσεις και αντιφάσεις και να γίνεται ε, όλο αυτό πριν και μέσα σε στοχευμένο πλαίσιο. Τελευταία μου παρατήρηση να πω τη δική μου γνώμη. Εγώ πιστεύω επίσης, τελευταία μου παρατήρηση, ότι υπάρχουν, ε, υπάρχει θέμα πόρων. Τα κονδύλια που έχουν προβλεφθεί είναι σημαντικά, αλλά δεν αρκούν. Αν δούμε τις διαστάσεις, για παράδειγμα, ε, του πρώτου κομματιού εκείνου του κεντρικού δικτύου ε, τουλάχιστον 250 δις <laughs> και ενώ υπάρχουν μόνο 31 δις προβλέπονται η διαφορά είναι τεράστια. Φυσικά θα πρέπει να γίνει και η ολοκλήρωση και από τα κράτη-μέλη. Αλλά νομίζω πως θα είναι απαραίτητο να αυξηθεί το κονδύλι ε, εξ αρχής. Αυτό ήθελα, αυτά ήθελα να πω αρχικά και στα υπόλοιπα θα επανέλθουμε. Well, thank you for that useful Ευχαριστούμε. Τώρα θα περάσουμε στην παρουσίαση της Κομισιόν και θα ακολουθήσουν ερωτήσεις από τους ε, σκιώδεις ε, εισηγητές. Κυρία Ιβάνοβα, Σμιτ, κυρία Ρίλε, Λανότε, Μπίλαν, τέσσερις σκιώδεις ηγητές και μετά κύριε Κοφεράτη θα λάβετε και εσείς ξανά τον λόγο. Ας περάσουμε τώρα στην εξολόγηση αντικτύπου του κυρίου Πακέ. Έχουμε τις διαφάνειές σας. Σας ε, καλωσορίζω λοιπόν. Παρουσιάστε μας την ε, πρότασή σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για τα σχόλιά του και χαίρομαι για την ευκαιρία που έχω να παρουσιάσω τα στοιχεία της αξιολόγησης αντικτύπου. Νομίζω πως θα ήθελα να σα παρουσιάσω τα των δύο ευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Έχουμε λοιπόν ένα από τα 12 μέσα που υπάρχουν. Οι υποδομές αυτές ε, θεωρούνταν πάντα η ραχοκοκαλιά της κοινή αγοράς και στις διάφορες προτάσεις της ε, Κομισιόν. και ευρύτερα στις στόχους ε, του 2020. Αυτό προκύπτει και από την ανάλυση της Κομισιόν και το 2030-2050 και η πολιτική αυτή είναι η βάση των υποδομών για την πολιτική των μεταφορών. Εάν δείτε την πολιτική αυτή προσπαθούμε να έχουμε μια προσέγγιση των επιτευγμάτων, των λαμπρών αυτής της πολιτικής των 15 ετών. Είχαμε πολλές επιτυχίες για τα βασικά έργα αυτά τα οποία όρισαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων τη δεκαετία του 90 έχουμε εμβληματικές επιτυχίες οι συνδέσεις ε, Βρυξελών, Λονδίνου, Παρισίων, Κολονίας ε, αλλά τώρα είναι και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και οι υποδομές αυτές ε, προσφέρουν αλλακτικέ για πολίτες και επιχειρήσεις. Τα βασικά προβλήματα χάραξης της ε, πολιτικής οφείλονται στο ότι βεβαίως πρόκειται για αρμοδιότητα κρατών μελών και ένωσης και στην πραγματικότητα τα περισσότερα από αυτά γίνονται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Το επίπεδο της Ένωσης συντονίζει και συνεισφέρει. Οπότε, σε τελική ανάλυση, προσφέρει ένα πλαίσιο στις εθνικές πολιτικές να συντονιστούν, να συντονίσουν το ευρωπαϊκό στοιχείο για να γίνουν οι εθνικές υποδομές και οι ευρωπαϊκές. Βεβαίως, το σύστημα αυτό τα προσφέρει αυτά Τέλεια και έχουμε περισσότερο ένα μοσαϊκό παρά ένα δίκτυο. Επίσης, έχουμε μία υποδομή ε, λιμάνια, αεροδρόμια, αλλά δεν συνδυάζονται αυτά στρατηγικά και εξαρτάται η υποδομή από τις τεχνικές προδιαγραφές στα εθνικά συστήματα υποδομών που εμποδίζουν μετά την ανάπτυξη ευρωπαϊκών ε, υπηρεσιών. Αυτό ειδικά στα τρένα ποιες είναι οι λύσεις. Να επικεντρωθούμε στο να πάμε από το μοσαϊκό, από την κουρελού αυτή σε ένα δίκτυο και να δούμε βεβαίως και κάποιες στενοπούς στα εθνικά δίκτυα που εμποδίζουν ε, τη λειτουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος να γίνει περισσότερο διατροπικό το δίκτυο, να δούμε την δυνατότητα συνδυασμού μέσων μεταφοράς, να γίνει διαλειτουργικό, να επιτρέψει στις εταιρείε να διατρέχουν εθνικά συστήματα μεταφορών, έξυπνες δηλαδή λύσεις που εφαρμόζονται σε όλα τα μέσα μεταφοράς και καλύτερη χρήση των υποδομών. Το η συγγήτρια πόσο δύσκολο είναι ο εισηγητής να δούμε πόσο σημαντικό είναι ε, να δημιουργηθούν οι νέες υποδομές και να δούμε και τις ανησυχίες των πολιτών. Γιατί όταν κατασκευάζεται η υποδομή βεβαίως επηρεάζει την περιοχή. Οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο μέγιστο την υφιστάμενη υποδομή και να κατασκευάζουμε νέα μόνο όταν είναι απόλυτος απαραίτητο. Και βεβαίως να διασφαλίσουμε πως το πρόγραμμα των διευρωπαϊκών δικτύων να είναι πιο αυστηρό στο πλαίσιο του. Για να στηρίξουμε λοιπόν την προετοιμασία της πρότασης βεβαίως κάναμε μια αξιολόγηση αντικτύπου. Υπήρχε μια αρκετά μεγάλη φάση διαβούλευσης, ε, πολύ μεγάλη ξεκινήσαμε το 2008 και πρόταση καταθέσαμε το 2011 μόλις. 3,5 ε, χρόνια λοιπόν από πλευρά υποψιών, ε, αλλά ήταν πάρα πολύ χρήσιμα αυτά ε, για να δούμε βεβαίως την άποψη όχι μόνο ε, αυτών οι οποίοι δρούσαν στο παρελθόν, τα κράτη-μέλη δηλαδή, αλλά και αυτών που συμμετέχουν στα έργα αυτά τον κλάδο, τις περιφέρειες, όσους επηρεάζονται από τα έργα αλλά και όσους τα χρησιμοποιούν. Και βεβαίως εκεί είχαμε κάποιες επιλογές. Υπήρχε πάντα επιλογή μηδέν όπως ε, γίνεται πάντα, δηλαδή το να μην αλλάξουμε την πολιτική. Ανέφερα ήδη αρκετά πράγματα. Και βεβαίως επηρεάζει τη λειτουργία της ε, κοινή αγοράς και υπάρχει και μια για τις περιφερειακές ε, περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, έλλειψη πρόσβαση στην κοινή ώρα. Έχουμε λοιπόν δύο επιλογές ε, πολιτικής και χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες νομίζω πως δεν έχουμε μεγάλες διαφορές. Έχουμε 25 πιθανές επιλογές αλλά τις φέραμε στις δύο. Η μία είναι κατ' ουσία να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με βάση τα υφιστάμενα έργα προτεραιότητας αυτά τα οποία έχουν ορίσει οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Υπάρχει Λιόν ε, Τωρίνο, υπάρχουν διάφοροι διάδρομοι, μεγάλα δηλαδή έργα. Ε, μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτά και να δούμε καλύτερα την εφαρμογή. Η άλλη επιλογή ήταν αυτή την οποία διατηρήσαμε να φύγουμε από τους μεγάλους άξονες και να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε με βάση μια ευρωπαϊκή μεθοδολογία ένα λεγόμενο δίκτυο πυρήνα με πιο εύρωστη ε, θα λέγαμε εφαρμογή. Αυτές τις δύο επιλογές συγκρίναμε. Ε, δεν ξέρω τώρα αν μπορείτε να τα διακρίνετε, αλλά σας τα έχω δώσει και σε φωτοτυπίες. Όταν συγκρίνουμε λοιπόν την επιλογή 1 και 2 νομίζω πως και οι δύο οπωσδήποτε αποτελούν βελτίωση η επιλογή 2 έχει θετικότερο οικονομικό αντίκτυπο λόγω του δικτύου αντί για μεμονωμένα έργα και βεβαίως λόγω της καλύτερης συνδεσιμότητας σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά βεβαίως υπάρχει και ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος και στις δύο περιπτώσεις η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του συστήματος βελτιώθηκε αλλά όσον αφορά τη χρήση γης, τη βιοπικιλότητα η επιλογή 2 έχει την επιλογή να χρησιμοποιεί την υφιστάμενη υποδομή περιορίζοντας έτσι τον αντίκτυπο αυτών. Αυτή είναι λίγο πολύ η διαδικασία που ακολουθήσαμε, που μας οδήγησε στην πρόταση της Κομισιόν του Οκτωβρίου 2011, που νομίζω πως έχει κάποια χαρακτηριστικά μπορώ να συνοψίσω σύντομα, αν μου επιτρέψετε, αν μου δώσετε στιγμή. Σας ευχαριστώ. Πρώτον, να προτείνουμε έναν κανονισμό για τα διευρωπαϊκά δίκτυα και όχι απόφαση, η ποιότητα βεβαίω ε, εξαρτάται από την ουσία, όχι από το μέσο, αλλά η απόφαση σήμερα απευθύνεται στα κράτη-μέλη, ε, που είναι οι βασικοί φορείς βεβαίω. αλλά αν επιλέξουμε κανονισμό έχουμε τη δυνατότητα να απευθυνθούμε σε όλους τους ενδιαφερόμενους στα λιμάνια, στις περιφέρειες σε όσους διαχειρίζονται τις σιδηροδρομικές υποδομές, όλοι μπορούν να συνεργαστούν. Δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό, έχουμε δύο στρώματα, το δίκτυο πυρήνα, το πιο ορατό κομμάτι βεβαίω, που αναπτύχθηκε με βάση μια ευρωπαϊκή μεθοδολογία, που θα μπορούμε να συζητήσουμε κάποια στιγμή αν σας ενδιαφέρει και στόχο έχει να συνδέσει και τα 27 κράτη-μέλη και μετά συνδέει τα κύρια ευρωπαϊκά λιμάνια, σημεία εισόδου και εξόδου και τα βασικά οικονομικά κέντρα της Ευρώπης. Οπότε φεύγουμε από μια προσέγγιση όπου έχουμε πρώτα το εθνικό δίκτυο και θέλουμε να το συνδέσουμε και πάμε σε μια ευρωπαϊκή μεθοδολογία. Το δίκτυο πυρήνας καλύπτει και τα 27 κρατημέλη με τρόπο ομοιογενή και έχουμε μετά το συνολικό δίκτυο που βασίζεται και στι εθνικές προτεραιότητες και στη διασύνδεση τους και τα δύο δίκτυα ε, έχουν την ίδια τις ίδιες προδιαγραφές αλλά η διαφορά είναι ότι το 2030 θα τελειώσει το ε, δίκτυο πυρήνας ενώ το άλλο το 2050. Και βεβαίω το δίκτυο πυρήνα είναι το απολύτω απαραίτητο, καθώ μιλάμε για πρόσβαση από όλε τι ευρωπαϊκέ περιφερείες μέσω αυτού του δικτύου στην εσωτερική αγορά. Και μετά η τρίτη πτυχή του ε, κανονισμού είναι, όπως είπα, να υπάρξουν ε, για όλα ε, τα μέσα μεταφοράς, ε, να υπάρξει διαλειτουργικότητα και οπωσδήποτε να δούμε και την ε, ποιότητα όσον αφορά ε, τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο όπως είπα πέρα από το πλαίσιο προγραμματισμού είχαμε και τα μέσα της εφαρμογής και εδώ πέρα έχουμε τρία μέσα που είναι σημαντικά τους βασικούς διαδρόμους που ανέφερε και ο εισηγητής βασιζόμαστε στην υφιστάμενη εμπειρία υπάρχουν ήδη δηλαδή ε, πολλά από αυτά είναι προτάσεις του Κοινοβουλίου δύο συντονιστές παραδείγματο χάρη είναι και ευρωβουλευτές και βοηθούν τα κράτη-μέλη και την Κομισιόν να εφαρμόσουν τις προτεραιότητες και θα ενισχυθεί η δουλειά τους και θα εστιαστούμε στους βασικούς αυτούς διαδρόμους που δεν είναι άλλο ένα επίπεδο προγραμματισμού ο προγραμματισμός είναι μόνο το δίκτυο αλλά υπάρχουν κάποια τμήματα από τα οποία είναι πιο δύσκολα εκπείρας το γνωρίζουμε αυτό και στα πιο δύσκολα αυτά κομμάτια προτείνουμε κάποιους διαδρόμους του κτηρίου πυρήνα για να δούμε καινοτόμες ε, χρηματοδοτικές λύσεις να Έχουμε συγχρονισμένη χρηματοδότηση μεταξύ κρατών μελών και εξίσου σημαντικό να φροντίσουμε να εμπλέκονται οι χρήστες στην βελτίωση των υποδομών. Βεβαίω, το τελευταίο εφαρμοστικό εργαλείο είναι κανονισμός, ε, δηλαδή το μέσο συνδέοντα την Ευρώπη, η ευρωπαϊκή συνεισφορά εδώ πέρα, που προτάθηκε ταυτόχρονα από την Κομισιόν με χρηματοδότηση 31,7 δισεκατομμυρίων ευρώ και ένας κατάλογος προκαθορισμένων έργων είναι δηλαδή αυτά στο δίκτυο πυρήνα που θα πρέπει να έχουν εφαρμοστεί μέχρι το 2020 και θα μας επιτρέψουν άρα να ξεκινήσει η ανάπτυξη του δικτύου αυτού ε, για να λειτουργεί το 2030. Τα έργα αυτά είναι αυτά με τη μέγιστη ε, προσθέμενη ευρωπαϊκή αξία, είναι διασυνοριακά, είναι στενοπή, είναι διατροπικά και διαλειτουργικά. for you to see it, but it's one of the δεν μπορείτε βεβαίω να τα διακρίνετε στο χάρτη. Ε, βλέπετε το, το σιδηρόδρομο εδώ πέρα, τα σιδηροδρομικά ε, και υπάρχουν τέσσερι, τέσσερις τέτοιοι χάρτες. Ο ένας αφορά επιβατικό δίκτυο σιδηροδρόμων, εμπορευματικό δίκτυο σιδηροδρόμων, και μετά έχουμε και οδικές μεταφορές και ποτάμιες. Καταλήγοντας λοιπόν κύριε Πρόεδρε, η πολιτική που προτείνει η Κομισιόν βασίζεται στο υφιστάμενο πλαίσιο Στόχο έχει λοιπόν η αξιολόγηση που να δει την ε, κινητικότητα αγαθών και ανθρώπων στην εσωτερική αγορά. Είναι ρεαλιστική και φιλόδοξη ταυτόχρονα. Ρεαλιστική υπό την έννοια πως χρησιμοποιεί στο μέτρο του δυνατού την υφιστάμενη υποδομή. Γιατί είναι και οι καιροί δύσκολοι Οπότε είναι ρεαλιστική αλλά και εστιασμένη και ταυτόχρονα είναι φιλόδοξη γιατί σημαίνει πως θα προωθήσουμε τη δέσμευση των κρατών μελών μέχρι το 2030 και είναι δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεισφέρουν σε ένα βασικό δίκτυο μέσω του προπολογισμού και βεβαίως μέσω και των μέσων εφαρμογής. Σας ευχαριστώ. Ε, μα, ε, λίγο. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Και βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Well, Ευχαριστούμε πάρα πολύ ο Πρόεδρος γιατί νομίζω ότι μας βοηθήσατε πάρα πολύ μας σε αυτά τα πλαίσια για κάτι που μας έχει απασχολήσει. Μας δώσατε κάποιες κατευθύνσεις και αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να μας δώσετε έναν τέτοιο χάρτη πάρα πολύ ωραίο, το βάλουμε στο γραφείο και να βλέπουμε πού είμαστε όσον αφορά το κορ. Κύριε Κοφεράτη, εσείς κάνετε την εισηγήσή σας. Μπάς και οι σκιώδεις έχουν κάτι πριν ξαναλάβετε το λόγο. Κύριε Βανόβο, ευχαριστώ πρόεδρε. Αναμφίβολα η ανάπτυξη αυτού του δικτύου είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό και για την εσωτερική αγορά και για την κινητικότητα επιβατών, εμπορευμάτων κλπ. Συμφωνώ με τα όσα είχε πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμφωνώ για τόσα είπε σε σχέση με τη βελτίωση του δικτύου και σε αυτή την αρχική φάση της ανταλλαγής των απόψεων θα σταθώ στα τρία βασικά. Καταναλωτής, εσωτερική αγορά, τεχνικά θέματα, τεχνοκρατικά θέματα και οικονομικά. Βέβαια, ο εισηγητή μα έδειξε κάποια από αυτά, οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν αναπτυχθεί αυτό το δίκτυο να μην έχουμε παραπάνω γραφειοκρατία. Να μην έτσι δημιουργηθεί φραγμό όσον αφορά την προσβασιμότητα του κόσμου. Ούτε να οδηγηθούμε σε όθηση των τιμών προ τα πάνω. Και το πάρα πολύ σημαντικό το οποίο ανέφερε και ο Σκοπεράτη ήταν το θέμα τη εναρμόνισης, αυτό το οποίο ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, τη διαγωνισμή για τα έργα υποδομής, διότι σίγουρα χρειάζεται να υπάρχει προσβασιμότητα στην πληροφορία όσον αφορά τις διασυνδέσεις, τη διαλειτουργικότητα σε σχέση με τα εθνικά δίκτυα και έτσι να έχουμε μια εύρυθμη λειτουργία του δικτύου για όφελος του επιβάτη και οπότε έτσι να μπορούμε να καλύψουμε κάθε είδος μεταφορά σε όλα τα κράτη-μέλη και να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε εισιτήρια τα οποία να καλύπτουν όλους τους τρόπους μεταφοράς. Reduced mobility, disabled passengers, uh, because there are still lots of disparities in, in different member states uh, related to these. Και να δούμε πώς θα εξομαλύνουμε, πώς θα λάβουμε υπόψη ε, τις διαφορές των κρατών μελών. και να δούμε τι θα γίνει εκεί που έχουμε κλιματικημένες περιοχές και να δούμε πώς είναι δυνατόν τελικά να πετύχουμε την, την, την ε, εκτέλεση των έργων ε, σε κάποιο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώ θα εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση και ο πολίτη, γιατί πάρα πολύ συχνά τα έργα, τα προγράμματα, τα projects καθυστερούν, γιατί έχουμε αντίθεση, αντίθεση δυναμική του, του, του, του κόσμου, των τοπικών κατοίκων ε, τόπιον. Οπότε ε, θα πρέπει να δούμε και για τα πιο επίμαχα από αυτά τα projects τι θα γίνει. Τώρα, όσον αφορά τι τεχνοκρατικέ πτυχέ του θέματο, ε, αναφέρεται το θέμα του ευρωπαϊκού συντονιστή, η δυνατότητα να εμπλαϊκεί ο συντονιστής με επιπλέον αρμοδιότητες και να δούμε πώς θα περιχαρακώσουμε το, το καθεστώς που θα διέπει τον ε, συντονιστή γιατί δεν πρόκειψε σαφώς ε, η διάρκεια της εντολής. Ε, νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει να ξεκαθαριστούν πριν αποφασίσουμε για τις αρμοδιότητες. Τώρα, το τελευταίο, όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά, συμφωνώ με τον εισηγητή μας. Όντως υπάρχει σπάνιση όσον αφορά τις, τους, τους πόρους, και επομένω, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκρινίσει το πώς βλέπει τον ρόλο της Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Μέχρι σήμερα η χρηματοδότηση προέρχεται από, από, από τα, τα, τα, μέσα συνοχής και διευκόλυνσης. Άρα, Επιτροπή, πώς βλέπετε ε, κάποια χείρα βοηθεία που το συμπίνουν για την ε, χρηματοδότηση των προγραμμάτων. Ευχαριστούμε κύριε Βάνοβα. Ο κύριο Όλε Σμιτ λαμβάνει τον λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο ε, Κοφεράτη αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρώτη μου ερώτηση ε, είναι κάπω ομή. Ο νέο κανονισμός θα πετύχει το στόχο του για αυτά τα δίκτυα. Θα βελτιώσει την κατάσταση. Διότι θα ήθελα πραγματικά να μου πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποια είναι η προστιθέμενη αξία από αυτόν τον οργανισμό. Θα έχουμε τη, κάποιο δυναμική βάση τόσο ώστε τα ευρωπαϊκά θεσμικά έργα να, να μπορούν να πούν στα κράτη-μέλη κάντε αυτό, κάντε εκείνο. Έχω ασχοληθεί σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο πάρα πολλά χρόνια σαν πολιτικό και Τώρα που βλέπω εδώ πέρα στην ε, σελίδα 3, εκεί που λέει ε, προγραμματισμό. προγραμματισμός, Α πούμε αυτό το ίδιο. Ο γεωγραφικό σχεδιασμό και προγραμματισμό είναι κάτι πάρα πολύ βασικό για τον κόσμο. Στην ε, Δανία προσπαθούμε να χτίσουμε ένα δρόμο και όλοι όσοι μένουν εκεί κοντά διαμαρτύρονται. Προσπαθούμε. Φτιάχνουμε ράγε για του οδρόμου και όλοι διαμαρτύρονται και λένε άντε φτιάχτε τούνελ. Προσπαθήσαμε να ληφθούν οι αποφάσεις όχι σε τοπικό αλλά σε περιφερειακό επίπεδο. Ε, αυτό ήταν αδύνατο. Γιατί υπάρχουν κάποια συμφέροντα τα λεγόμενα εθνικά συμφέροντα που ίσως το κοινοβούλιο, ίσως η κυβέρνηση είναι καλύτερα να τα κάνει. Πολύ δύσκολα. Δεν θέλω να τα περιπλέξω περισσότερο τα θέματα, αλλά σας ερωτώ. Τα σκεφτήκατε. Αυτό είναι η πρώτη μου ερώτηση. Τώρα, δεύτερη ερώτηση. Για τη χρηματοδότηση. Έλα, ναι. Θα μας δώσει αυτό περισσότερα χρήματα για τα, για τα έργα γιατί μας λείπουν λεφτά, όπως είπατε και εσείς κύριε Γοφεράτη. Είμαστε και στην Επιτροπή Κρίσης και εκεί το βλέπουμε πολύ ξεκάθαρα. Third question. Because that is of... Και η τρίτη μου ερώτηση, γιατί φυσικά η χρηματοδότηση αφορά τα μέλη τα κράτη-μέλη. Γιατί αν τα κράτη-μέλη μπορεί να λένε ναι, ναι, η Ευρώπη να τα χρηματοδοτήσει αυτά, αλλά εμεί λεφτά γιοκ. Και αν θέλουμε όντω να ενωθεί, να συνδεθεί η Ευρώπη, γιατί περί αυτού πρόκειται, Εάν δεν υπάρχουν οι συνδέσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη, μπορεί να έχουμε κάποιε διασημερινοριακές συνδέσει, αλλά μετά τίποτα άλλο. Λέμε και εκείνη τη γέφυρα στη Δανία, αλλά όταν την περάσει κανείς εκείνη υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα πιο μέσα στη Δανία. Και έπειτα αυτό το θέμα με τον Ευρωπαίο συντονιστή. Τι είναι αυτός και τι είδος εντολή θα έχουν αυτοί οι συντονιστές. Και πώς θα επιβάλλουν τους κανονισμούς ή τις αποφάσεις μας στα κράτη-μέλη. Πολύ θα ήθελα να ακούσω την απάντησή σας, κυρία μου. Και η τέταρτη μου ερώτηση είναι η εξή. Εγώ ξέρω ότι τα φορτηγά τρένα κατά μέσο όρο τρέχουν με 30 χιλιόμετρα την ώρα. 30, ναι, όλα και όλα. Ποια είναι η μέση ταχύτητα ενός φορτηγού τρένου που πάει από τα ορυχεία πάνω στα βορεινά της χώρας μου μέχρι τα ναυπηγεία στην Ισπανία. Πόσες μέρες κάνει και ποια είναι η μέση ταχύτητα. Αυτό μου είπαν εμένα πριν από δύο χρόνια. Συγγνώμη, όχι 30, 13. 13 χιλιόμετρα. Σχεδόν αδύνατο είναι. Άρα θα πρέπει να αλλάξετε τα τρένα και ε, η διαλειτουργικότητα επομένως δεν ευωδώνεται. Επομένω, κύριε Χάρβορτ, να σα πω ότι 100% μόνο την καρδιά συμφωνώ με αυτό, όμω διατηρώ κάποιε αμφιβολίε. σω χρειαζόμαστε κάποια πιο αποφασιστικά δυναμικά μέτρα. Χάρβορτ, ευχαριστούμε για τι ερωτήσει που πάντοτε είναι κρυστάλλινε. Έχουμε επομένω τώρα του υπολείπου ε, σκιώδηδε, ε, Μπίλεν, Μπαχίαν. Ε, Όποιο θέλει τέλο πάντων μπορεί να λάβει το λόγο. Καλό είναι το ότι μιλάω αμέσως με τον κύριο Σμιτ γιατί μίλησε πως υπάρχουν διαφορετικά κόμματα και διαφορετικές απόψεις. Στην πόλη μου, στη Στουτγκάρδη, ξέρετε πως γίνεται χαμός ακριβώς για τα προβλήματα τα οποία αναφέρατε. Ε, αν πάει η Κομισιόν Στουτγκάρδη με μια διαδικασία επί παραβάση, ή επιβάλλει ή ζητήσει να χτιστεί γρήγορα το έργο θα είναι ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα και είναι ενδιαφέρον. Νομίζω πρέπει να σκεφτείτε κύριε Κονφεράτη πως ε, μπορούν να έχουν ένα ρόλο επίλυσης ε, διαφορών ε, οι συντονιστές. Χρειάζεται αυτό για μεγάλα έργα υποδομών γιατί βεβαίως οι πολίτες δικαίως αναρωτιούνται αν έχουν νόημα αυτά τα έργα, αν είναι τα σωστά έργα για τα χρήματά τους. Αυτό έγινε στη Στουτγκάρδη αν χρησιμοποιούνται σωστά τα χρήματα των φορολογουμένων ή μήπως μπορούσε να κατασκευαστεί αλλιώς το μεγάλο έργο το Στουτγκάρδι 21 που λέγαμε. Καλό ήταν λοιπόν η Κομισιόν να τα σκεφτεί αυτά γιατί βεβαίω ε, μιλάει και θα πρέπει να συνεργαστεί με περιφέρειες, ε, κράτη, μέλη, είναι μεικτά τα έργα, μεικτή η ευθύνη, οπότε καλό είναι εκ των προτέρων να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε επίλυση διαφόρων. Το ένα είναι αυτό που ήθελα να πω και ήθελα να στηρίξω και τον συγητή και πρέπει να ορίσουμε τον ρόλο των συντονιστών αλλά μια διεύρυνση νομίζω θα μπορούσε να οδηγήσει και σε συγκεκριμένη συνεισφορά της Επιτροπής μας. Κάτι άλλο θα ήθελα να αναφέρω. Μιλήσατε για τα οικονομικά και συμφωνώ. Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα όσον αφορά τα οικονομικά. Εάν δείτε τα μεγάλα έργα και τις προκηρύξεις τους, θα δείτε πως κοστίζουν κατά κανόνα το διπλό από τον προϋπολογισμό τους. Οι δε προκηρύξεις δεν ε, λειτουργούν. Αυτό το πρόβλημα έχουμε με τα μεγάλα έργα, τα κατασκευαστικά το κόστος είναι διπλό αν όχι και μεγαλύτερο. Τότε πρώτα απ' όλα πρέπει να αναγράφεται το σωστό κόστος και να υπάρξει και μείωσή του αλλά και ευθύς εξ αρχής το κράτος και ο εργολάβος επιτέλους να, να πληρώνει κάποιους ε, όταν υπάρχουν τέτοιες υπερβάσεις. Πρέπει και εδώ πέρα δώσουμε βάρος. Κύριε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Κοφεράτη και τον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Μας έκανε πάρα πολύ αξιολογική εισήγηση και θέλω να σας πω ότι συμφωνώ με τον τρόπο με τον οποίο μας ε, ε, δώσατε το, το, το περίγραμμα των προβλημάτων ε, που μας εξηγήσατε τι ισχύει σήμερα σαν δίκτυα. Όντω ε, είναι κάτι, τώρα δεν έχουμε δίκτυο, έχουμε κάτι σαν <laughs> ψηφιδωτό και τέλο πάντων ε, θα πρέπει να υπάρχει, να υπάρξει ολοκλήρωση, ενοποίηση, είπαμε δεν έχουμε διαλειτουργικότητα και αυτό αφορά όλους τους τρόπους μεταφορών. Και πάρα πολύ με εντυπωσίασε πάντω ε, αυτό ο συγκριτικό πίνακα, αυτή η σύγκριση που έχετε στην σελίδα 11 τη μελέτη επιπτώσεων, εκεί που συγκρίνεται του, του, του, του, του πόρου που έχουν επενδυθεί εις ε, τη συνδρομική σύνδεση του Ίγκολσταντ. Ε, αυτά τα 25 λεπτά επίσης μα τα περιγράψατε, τα οποία, ε, τα οποία χάνονται στην διάβαση των συνόρων ε, οπότε αυτό είναι κακό για επιβάτες και για εμπορεύματα. Και επίση το πώς εξαρτώνται όλα από τον έλεγχο που γίνεται ή στο Μόναχο. Όλα αυτά δείχνουν ότι η κατάσταση επιδέχεται σημαντική βελτίωση. Εγώ προέρχομαι από ένα κράτος μέλος το οποίο όντω είναι πάρα πολύ πίσω όσον αφορά τι μεταφορέ. Είμαι Πολωνός και γι' αυτό σας λέω το θέμα αυτό με συναρπάζει. Όντω, υπάρχουν κάποια θέματα, και κάποια προβλήματα και το βασικότερο είναι το οικονομικό. Βεβαίως ισχύει ότι το έγγραφο αυτό το οποίο μας παρουσιάσατε μα οδηγεί να προτιμήσουμε την επιλογή υπαριθμών 2. Παρ' όλα αυτά, είναι η πιο ακριβή επιλογή. Μιλούμε για παραπάνω 15 δι που θα πρέπει να καλυφθούν από τι επόμενε δημοσιονομικέ προοπτικέ και γι' αυτό και θέλω να σα ρωτήσω το εξή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώ θα εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση σε σχέση τουλάχιστον με την δεύτερη επιλογή. Επίσης, έρχομαι να συμφωνήσω με τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι ε, μίλησαν για το ότι εδώ υπάρχει ο κίνδυνος να αυξηθεί η γραφειοκρατία. Για τις επιπλέον αρμοδιότητες του συντονιστού. Πώς θα εξασφαλίσετε. Πώς θα εξασφαλίσετε ότι η γραφειοκρατία δεν θα εμποδίσει την πρόοδο των έργων και προγραμμάτων. Τι θα γίνει επίσης και με την προστασία του περιβάλλοντος. Η κυρία Ρίλε μας είπε για αυτό το περίφημο θέμα του σταθμού της Στουτγάρδης. Στην Πολωνία, ξέρετε, έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις όσον αφορά τον διάδρομο που πάει από τη Βαλτική στην Νότιο Ευρώπη. Και έχουμε ένα σωρό διαμαρτυρίες ε, σε σχέση με τις περιοχές ε, του Natura 2000. Άρα, προσοχή, και στην Ανατολική Ευρώπη θα υπάρξουν σημαντικά προβλήματα. Ξέρετε, εκεί αρχίζουμε από το α, από το 0. Προσοχή επομένω και στην κοινωνική πτυχή του θέματο. Πιέζει ο χρόνο σήμερα το πρωί, αλλά βέβαια ο κ. Κοφεράτη όταν έρθει η ώρα θα το ξανασυζητήσουμε το θέμα. Μπαλτασάρι, Βερχάγεν. Παρακαλώ να είσαστε σύντομοι. Sorry, it's next. Sì, grazie Presidente. Sarò Μάλιστα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα γίνεται πιο σύντομος. Ευχαριστώ φυσικά τον Σέρτζο Κομφεράτη, καθώς και τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Βρίσκω πως αυτός ο προγραμματισμός είναι απαραίτητος ε, τόσο για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, όσο και ως μορφή επένδυσης και άρα ανάπτυξης, ε, την οποία χρειάζεται ε, οπωσδήποτε η Ευρώπη και η η μορφή, πιστεύω, του συντονιστή, των συντονιστών είναι μια κεντρική φιγούρα όσον αφορά τη δυνατότητα διαμεσαλάβησης που καλείται να κάνει και να, έτσι ώστε να συνδυαστούν οι διάφορες απαιτήσει τοπικές, περιφερειακές και κρατικές αλλά και ως υπεύθυνο μιας, ενός, ε, της υλοποίησης των έργων. Αυτό το νέο δίκτυο με, μεταφορών θα πρέπει να λάβει υπόψη και τις εξελίξεις που υπήρξαν ε, όσον αφορά τα γεωοικονομικά δεδομένα. Η Μεσόγειος είναι κεντρική σημασία. Στο 1 τρίτο του παγκόσμιου, της παγκόσμιας κίνησης σκαφών ε, περνά από τη Μεσόγειο. Όλα τα αγαθά που περνάνε έρχονται από την ε, Βραζιλία, από την Ινδία, από την Κίνα, περνάνε από το κανάλι του Σουέζ. <coughs> Οπότε φυσικά υπάρχει ανάγκη να ενισχυθούν τα δίκτυα και να αξιοποιηθούν ώστε να μπορεί κανείς να φτάνει γρήγορα και ασφαλώς στο κέντρο της Ευρώπης. Στον χάρτη υπάρχει όμως μια λευκή τρύπα και αυτή την ερώτηση θέλω να κάνω στην Επιτροπή που είναι τα Βαλκάνια. Μόλις χαιρετήσαμε τον εκπρόσωπο της Κροατίας που θα μπει πολύ σύντομα ως πλήρες μέρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα επόμενα χρόνια θα μπει και η Σερβία και οι άλλες χώρες των Βαλκανίων. Θεωρώ λοιπόν πως ένα συνολικό πρόγραμμα τέτοιου Ελληνικού δεν μπορεί μπορεί να μην συμπεριλαμβάνει και ένα σχέδιο για τα Βαλκάνια. Δεδομένου ότι το διάδρομο 8 που υπήρχε εκ των προτέρων έχει μείνει απ' έξω. Τέλος, το δημοσιονομικό πλαίσιο. 31 δις ε, ευρώ που προβλέπονται. 20 από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 10 από τα Ταμεία Συνοχής. Στην ουσία απευθύνονται στην ε, ολοκλήρωση των έργων ε, του τελευταίου, του τελευταίου μιλίου όπως λέγονται, δηλαδή αυτά που συνδέουν ε, μικρές παρεμβάσεις που συνδέουν ας πούμε το αεροδρόμιο με το κοντινό λιμάνι ενώ πρόκειται για τεράστια πρόγραμμα και μιλάμε για 1,5-3 Άρα καταλαβαίνετε το χάσμα είναι τεράστιο. Η Κομισιόν το έχει λάβει αυτό σοβαρά υπόψη. Αυτά τα project bond, τα ομόλογα έργου τα έχει λάβει σοβαρά υπόψη για αυτόν τον προγραμματισμό και για αυτά τα έργα. Για διαφορετικά μπορεί να μείνουν όλα αυτά επί χάρτου και πολύ δύσκολα τα κράτη θα μπορέσουν ε, χωρίς αυτό το μέσο χρηματοδότησης να έχουν την δύναμη τα χρήματα για να ε, υλοποιήσουν όλα αυτά τα προγράμματα διεθνή, υπερεθνικά. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να συμφωνήσω με αυτό το οποίο είπε ο για του συντονιστέ και το συντονισμό διαφόρων Εγώ είμαι σε μεθοριακή περιοχή και συζητάνε εκεί πέρα για τον Σιδερένιο Ρήνο, σύνδεση με τον Ντουίσμπουργκ που δεν προχώρησε γιατί υπήρχαν βεβαίως συγκρουόμενα συμφέροντα, εθνικά συμφέροντα για ένα έργο που θα ήταν τριεθνές. Όταν υπάρχει τέτοια κατάσταση είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Όταν ένα κράτος μέλος ε, θέλει να, να κάνει κάτι τέτοιο. Ποιο συμφέρον θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Γιατί να χρηματοδοτηθούν τέτοια έργα. Εκεί όπου υπάρχει πανευρωπαϊκό συμφέρον για βελτίωση των διασυνοριακών δικτύων των συνδέσεων μεταξύ διαφόρων γραμμών να έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση από ό,τι στο παρελθόν. Και άρα το πρόγραμμα συνολικά χρειάζεται περισσότερα κονδύλια. Γιατί ε, μα δείτε αν ασχοληθούμε μόνο με τα μεγάλα έργα σε πολλά κράτη-μέλη θα σταματήσουν τα έργα γιατί δεν υπάρχει χρηματοδότηση ή αλλού σε άλλα αν δεν αποτελεί πρώτη προτεραιότητα το συγκεκριμένο έργο, πάλι θα μείνει εκτός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα σχόλιο και από μένα. Νομίζω πως το όλο ζήτημα της διαλειτουργικότητας και των προδιαγραφών είναι οπωσδήποτε μεγάλο σημαντικό ζήτημα κατά μήκος ενός διαδρόμου και ξέρω πως οπωσδήποτε και ο Μπράιν Σίμψον της Επιτροπής Μεταφορών είναι απογοητευμένο από την έλλειψη προσοχής για τις αρχές ενιαίας αγοράς και από πλευράς τεχνικών κανονισμών, αμοιβαίας αναγνώρισης, διαλειτουργικότητας, όλα αυτά τα ζητήματα. Αλλά ε, ε, τα γνωρούμε αυτά συνεχώς στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σιδηροδρόμων Εδώ πέρα λοιπόν θα μπορούσε η Επιτροπή μας να ενισχύσει την Επιτροπή Μεταφορών. Δώσω το λόγο πρώτα στην Κομισιόν και μετά σε σας κύριε Κοφεράτη. Συμφωνείτε? Ωραία. Κύριε Πέκε, έχετε λίγα λεπτά να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Τόσα πολλά ακούστηκαν. Θα προσπαθήσω να δώσω κάποιες απαντήσεις, αλλά μάλλον θα πρέπει να κάνουμε και διμερείς συναντήσεις με τα μέλη που ενδιαφέρονται γιατί θα είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες για το γεωγραφικό θέμα. Το θέμα της προσβασιμότητας καλύπτεται από τις κατευθυντήριες γραμμές. Το άρθρο 43 είναι ένα θέμα κλειδί και επίσης ε, η έκδοση εισιτηρίων διατροπικών λοιπά, Όλα αυτά συμπληρώνουν άλλες ε, πολιτικές πρωτοβουλίες και άλλα αριθμιστικά πλαίσια και αποτέλεσαν τμήμα της συζήτησης κατά την ε, προετοιμασία και είναι μέρος της πρότασης όσον αφορά το ρόλο των συντονιστών και διαμεσολαβητών. Πώς γίνεται η εφαρμογή και η εγκατάσταση, μάλλον η κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής. Φυσικά είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο ε, όσον αφορά την πολιτική και όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και το τρόπος που θα αντιμετωπίσουμε το θέμα είναι να δούμε ε, τα ευθύνε ε, του κάθε επίπεδου διακυβέρνησης και έπειτα να προετοιμάσουμε και να συζητήσουμε το πρόγραμμα με τους πολίτες, το οποίο παραμένει στην εθνική ευθύνη ε, και εμείς δεν νομίζουμε ότι θα πρέπει αυτό να έρθει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν θα λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Ταυτόχρονα πρέπει να ε, θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν θέματα επικοινωνίας τα οποία δεν χειριζόμαστε πάντοτε σωστά. έχουμε περιπτώσεις όπου ε, το Μπρεν, όπως τον Μπρέναρο για παράδειγμα όπου ο μακαρίτης ε, Καρλ Φαν και τώρα ο Πατ Κόξ ε, είναι πολύ πιο αναμειγμένοι μετά από αίτημα των αρχών. Οι συντονιστές δηλαδή θα μπορούσαν να παίξουν το ρόλο της διάδοσης καλύτερης πρακτικής στην προπαρασκευή αλλά και να, δείξουν, να διαβεβαιώσουν, να εξασφαλίσουν μάλλον θα συνεχίζεται η επικοινωνία γιατί το θέμα ήταν να πιστούν και οι πολίτες ότι από τη στιγμή που προετοιμάζει κανείς το έργο και αρχίζει τη διαβούλευση και τη στιγμή που αρχίζει το, η κατασκευή υπάρχει ένα χρονικό διάστημα μεγάλο που δεν γίνεται καμιά επικοινωνία και όταν ξαφνικά αρχίζουν τα έργα ο κόσμος έχει ξεχάσει την αρχική εικόνα και ιδέα. Ο συντηνιστής ήδη παίζει το ρόλο του διευκολυντή και ίσως θα μπορούσε και να ενισχυθεί. Ο ρόλο του πάντοτε με σεβασμό στο γεγονό ότι σύμφωνα με την ε, συνθήκη η ευθύνη εφαρμογή του προγράμματο, του έργου, ε, βαρύνει τα κρατημέλη και δεν μπορεί να μετακινηθεί σε επίπεδο ένωση. Και έπειτα για το ρόλο των συντονιστών και για την έννοια ότι θα πρέπει να αποφευχθεί η γραφειοκρατία. Αυτό είναι σαφές. Πιστεύω πως ο αντίκτυπος είναι ακριβώς να διευκολύνει και να μπορέσουν έτσι τα έργα να γίνουν πιο αποτελεσματικά και πιο γρήγορα. Από αυτή την άποψη δεν νομίζω πως υπάρχει ανησυχία στα κράτη-μέλη για τη γραφειοκρατία, αλλά να εξασφαλίσουν ότι θα μείνουν υπεύθυνα για την εφαρμογή. Και αυτό δεν έχει αλλάξει, δεν έχει μετακινηθεί προς τον ε, συντονιστή. Εδώ το θέμα δεν είναι μόνο οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε πολιτικό επίπεδο, αντικατοπτρίζουν ε, τις ε, πολιτικές ε, προτεραιότητες, προτεραιότητες και προγράμματα έτσι ώστε η εφαρμογή να είναι πιο εύκολη αλλά και ο τρόπος με τον οποίο διατυπώνεται το νομικό κείμενο και οι νομικές διατάξεις ε, φαντάζομαι πως θα προκαλέσει η συζήτηση ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο γιατί το κείμενο έχει αναθεωρηθεί στο Συμβούλιο Μεταφορών για να δημιουργηθεί περισσότερη ευελιξία ε, αλλά είχαμε μια γενική προσέγγιση ε, λογική στις 23 Μαρτίου. Πάντως, ε, Πιστεύουμε ότι μέσω του κειμένου πρέπει, ε, προβλέπεται δέσμευση σοβαρή από τα κράτη-μέλη. Τελευταίο σημείο, ακόμα και αν ε, η χρηματοδότηση δεν είναι μέρος των κατευθυντηρίων γραμμών, μιλήσατε για περισσότερη ανάγκη χρηματοδότησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, κρατών μελών. Πρόκειται για ευρωπαϊκό δίκτυο, είναι ευρωπαϊκές οι προτεραιότητε, είναι ρεαλιστικό στην χρήση των υφιστάμενων υποδομών και τα διάφορα μέσα που προέρχονται, όπως οι διάδρομοι, προβλέπουν την επαρκή προετοιμασία ώστε να έχουμε καλύτερα προγράμματα. Και μόνο έτσι Ε, νομίζω ότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε όντως καλύτερη, ε, καλύτερο προγραμματισμό. Εάν τα κράτη-μέλη δεν έχουν σημαντικό προϋπολογισμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δύσκολα προγραμματίζουν και εκείνα, γι' αυτό και θα πρέπει να γίνουν διαπραγματεύσεις σχετικά στο επόμενο πολιετές, ε, αλλά και να έχουμε καλύτερα προγράμματα, καλύτερη προετοιμασία των προγραμμάτων, να κινητοποιηθούν και η Ευρωπαϊκή ε, Τράπεζα Επενδύσεων, χρηματοδότηση εθνική, ευρωπαϊκή και ρόλο των διαφόρων χρηματοδοτών. και η εργασία που γίνεται επί των προγραμμάτων, επί των, αυτών των προγραμμάτων θα παίξει ρόλο για τη χρηματοδότηση. Φυσικά δεν έχουμε ε, μαγική λύση ε, όσον αφορά τη χρηματοδότηση, αλλά πιστεύουμε πως ε, η πρόταση θα διευκολύνει διάφορα προγράμματα και ούτως ή άλλως θα εστιάσουμε την προσοχή στην υπάρχουσα, στις υπάρχουσες υποδομές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Όντως ε, πιστεύω πως οι βουλευτές θα θελήσουν να έρθουν σε διμερή επαφή μαζί σας. Ε, κύριε Κοφεράτη, τώρα ήδη τρώμε το χρόνο σας από το επόμενο σημείο. <laughs> Θέλετε να ολοκληρώσετε λοιπόν αυτή τη συζήτηση και να πείτε και για το χρονοδιάγραμμα. Ναι, θα είμαι πολύ σύντομο. Θέλω να ευχαριστήσω του συναδέλφου που με τα ερωτήματά του υπέδειξαν σημεία ενδιαφέροντα που θα παίξουν χρήσιμο ρόλο στην σύνταξη τη πρόταση. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Πακέ που ολοκλήρωσε την εισήγησή του με, με, κάτι το οποίο συμμερίζομαι. Το ίδιο το πρόγραμμα έχει μια μεγάλη δόση, περιλαμβάνει μεγάλη δόση ρεαλισμού αλλά και φιλοδοξία. Ρεαλισμό σε σχέση με το κόστο, γιατί το να ενεργήσουμε με βάση τα όσα υπάρχουν περιορίζει το κόστος. Ήθελα όμως να υπογραμμίσω και το θέμα της φιλοδοξίας. Εγώ επιμένω και ζητώ βοήθεια από όλους. Το πιο λεπτό θέμα είναι ότι πρόκειται για πολύ μεγάλη παρέμβαση Το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι η απαραίτητη συνένεση για την υλοποίηση τέτοιων μεγάλων έργων. Ξέρετε ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα ε, στους ε, αιρετούς εκπροσώπους και τους υπολείπους. Σπανίως ε, μπορούμε να εκτιμήσουμε τα αισθήματα των, των πολιτών. Γι' αυτό και πρέπει να δουλέψουμε πάνω στην γνώση και την συμμετοχή των ε, ανθρώπων ώστε να μπορέσουμε να δούμε, να διορθώσουμε αν δεν γίνεται και από την άλλη πλευρά να μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις. Εγώ εδώ λοιπόν πιστεύω και ελπίζω πολύ στη συνεργασία με τους συναδέλφους και επειδή το πιστεύω θα έχουμε την ευκαιρία να το ξανασυζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που αναλάβατε αυτή τη σημαντική έκθεση. Θα στείλετε λοιπόν ένα σχέδιο έκθεσης στις 30 Μαΐου και 20-21 Ιουνίου θα το εξετάσουμε, τροπολογίες ε, τον Ιούλιο, 10 Ιουλίου και υιοθέτηση στη... τον Οκτώβριο για την ε, Επιτροπή Μεταφορών. Κάποιος είπε ότι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε και στις δύο επιτροπές και σίγουρα η Επιτροπή Μεταφορών θα μας ε, βοηθήσει. Περνάμε στο επόμενο θέμα τώρα. Θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Κλένκοβιτς από την Κροατία που επίσης σήμερα ήρθε για πρώτη φορά. Έχετε αυτή τη ροζ κάρτα για τους παρατηρητές. Αν και δεν έχουμε κάποιον ε, συγκεκριμένα στην Επιτροπή μας, εμείς σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Και περνάμε τώρα στη δεύτερη έκθεση του κ. Κοφεράτη. Πολύ σκληρά δουλεύει ο κ. Κοφεράτη. και μια γνωμοδότηση τη Επιτροπή Απασχόληση για το Λευκό Βιβλίο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια ατζέντα για επαρκή και βιώσιμε συντάξει. Η κυρία Όμεν Ρόιτεν είναι η συγκίτρια στην Επιτροπή Απασχόληση. Έχουμε σκιώδης εδώ, δεν είμαι βέβαιο αν πρέπει να... Ποιο είναι από το ΕΛΚ, ε, η κυρία Χάνσλικ, μάλιστα. Ο κύριο Κρόιτσμαν, μάλλον Μάντερ. μιλάει για του φιλελεύθερους, Τούρνεν δεν είναι εδώ. Εγώ εξομονόματος στο ECR. Ο κύριο Ντιγιόγκ είναι εδώ επίση τον καλωσορίζω. Κύριε Κοφεράτη, θα μας πείτε την εκτίμησή σα, Δεν έχουμε και πολύ χρόνο, αλλά ας ξεκινήσουμε. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η σημασία του θέματος αυτού είναι γνωστό. Του θέματος των συντάξεων είναι γνωστό. Δεν χρειάζεται να μακρηγορήσω για αυτό το θέμα. Το γεγονός ότι η Κομισιόν έφτιαξε και λευκό βιβλίο παραδεικνύει ότι ε, είναι μεγάλες οι συνέπειες για την Ευρώπη και τα προβλήματα είναι αυτά που δείχνει και ο τίτλος. Δεν είναι μια περίπτωση, δεν είναι τυχαίο που χρησιμοποιήσαμε τα λέξη, τις λέξεις ε, συντάξεις κατάλληλες, ασφαλείς και βιώσιμες. Ο κύκλος αντιδράσης της οικονομίας με την κρίση που διανύουμε ε, έθεσε υποσυζήτηση την ε, αντοχή αυτών των συστημάτων προνοίας και ταυτόχρονα και τις ανάγκες των ανθρώπων που χρειάζονται αυτά τα συστήματα προνοίας. Γι' αυτό θέλουμε να εναρμονίσουμε και τα ε, συντάξεις για τις διάφορες χώρες που διαφέρουν ε, για λόγους όπως οι μεταφορές αλλά και η κοινωνική συνοχή που Ταυτόχρονα μαζί με την ε, εναρμόνιση θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι απαραίτητες μάλλον ε, ε, διασφαλίσεις για την κάθε διάταξη. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να εντοπίσουμε ποια είναι τα βασικά προβλήματα για να υπάρξει σταθερότητα. Είναι απαραίτητο να φτάσουμε σύντομα να, στην ευθυγράμμιση της, συνταξι, της ηλικίας σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και να συνδεθεί η ηλικία αυτή με την αύξηση της ε, του προσδόκιμου βίου. Γιατί η οικονομία υπόκειται τις ε, επιπτώσεις της κρίσης. Ε, γι' αυτό το λόγο πιστεύω πως είναι απαραίτητο για να υπάρξει σταθερότητα σε συστήματα, να φτάσουμε σε μια ευθυγράμμιση της, της ηλικίας συνταξιδότησης για τους άντρες και για τις γυναίκες, αλλά ταυτόχρονα η, η αύξηση της, της ηλικίας συνταξιδότησης να ήταν σκόπιμο να συνδεθεί με εθελοντική, εθελούσια ε, συνταξιδότηση μέσω ενός συστήματος κινήτρων ε, για να μπορούν να εργάζονται περισσότερο τα άτομα, αλλά, αν το επιθυμούν, αλλά χωρίς δεσμεύσει που μπορεί να είναι αντιπαραγωγικές για το σύστημα στο σύνολό του ή για τα μεμονωμένα εθνικά συστήματα. Στη διάρκεια αυτών των ετών αυξήθηκε και ο αριθμός των ατόμων που εγκατέλειψαν την εργασία τους πριν από την προβλεπόμενη ε, ηλικία. Ε, κρίση, λόγω της κρίσης στο μεταπητικό τομέα αλλά και στις υπηρεσίες. Χρειάζεται αυτό να περιοριστεί, αλλά για να περιοριστεί θα πρέπει να υπάρχει μια αναπτυσσόμενη οικονομία που θα, θα δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης και ε, ταυτόχρονα να υπάρχει παράλληλα ένα είδος προστασίας εγγυημένης με την απαραίτητη ε, στήριξη όσον αφορά την συμβολή των ανθρώπων. Είδαμε τα τελευταία χρόνια ότι και λόγω αντικειμενικών απαιτήσεων δίνεται προτεραιότητα σε ένα σύστημα το οποίο θα έχει τη δυνατότητα την κεφαλοποίηση, δηλαδή την καταβολή των συμβολών ως εφάπαξ. Ε, ε, αυτό αρχίζει να υπερισχύει, όμως η καταβολή ε, των ενισχύσεων των, ε, μάλλον των ε, συμβολών. Αυτό σημαίνει περισσότερα κατακαιρματισμένη εργασιακή ζωή και γι' αυτό θα πρέπει να ε, στηριχθεί κανείς από συμπληρωματική επικουρική σύνταξη, από το δεύτερο πυλώνο δηλαδή είναι ένα σημαντικό στοιχείο του Λευκού Βιβλίου, αλλά ίσως και να είναι και το πιο σημαντικό στοιχείο που εμείς θα θα πρέπει να απασχολήσει. Γιατί είναι απαραίτητο να εντοπίσουμε λύσεις που δίνουν εξασφαλίσει για τις επενδύσεις που εγγυώνται τα κεφάλαια που θα χρησιμοποιηθεί στο τέλος και για την επικουρική σύνταξη, δηλαδή για το δεύτερο πυλώνα. Να θυμίσω ότι όσον αφορά την διαδικασία, την σταδιακή και την αναρμονική ε, αύξηση της ηλικία δεξιδότηση υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορά τις γυναίκες. Η εξίσωση της ηλικία δεξιδότηση για τις γυναίκες με αυτή της, ε, των ανδρών είναι απαραίτητη, αλλά δεν μπορούμε να ξεχνάμε πως οι γυναίκες έχουν μια ε, δραστηριότητα μεγαλύτερη γιατί συνήθως αυτοί, αυτές είναι που αναλαμβάνουν τη φροντίδα παιδιών και συζύγου. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εισαχθούν λύσεις που θα μπορούν να αναγνωρίσουν αυτές τις ε, υπηρεσίες φροντίδας ή την διακοπή της επαγγελματικής σταδιοδρομίας την οποία αναγκάζονται να κάνουν οι γυναίκες πιο συστηματικά λόγω της μητρότητας. Είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του γυναικείου φίλου, όσο το κάνουμε. Η φροντίδα μπορεί να τη μοιραστούν, αλλά τη μητρότητα όχι. Άρα λοιπόν όλα αυτά θα πρέπει να μπουν μέσα στις ε, διατάξεις αλλά και να εισαφθούν τα στοιχεία που θα επιτρέψουν την ενίσχυση όσον αφορά της δημόσιας πρόνοιας αλλά και την βεβαιότητα περί της τελικής χρήσης όσον αφορά την ε, επικουρική σύνταξη, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι σε αυτή την περίπτωση έχουμε νέα προβλήματα που χαρακτηρίζουν την ε, δυνατότητα κυκλοφορίας, ελεύθερης κυκλοφορίας των ατόμων. Δηλαδή, δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων αλλά και εναρμόνιση των κριτηρίων και των φορολογικών κριτηρίων που αφορούν το σύνολο των πόρων που επενδύονται για την επικουρική σύνταξη αλλά και πιο συγκεκριμένα λύσεις ε, λεπτομερείς σε σχέση με αυτήν την επικουρική σύνταξη. Δηλαδή, πρόνοια δημόσια αλλά συνδεδεμένη και με το δεύτερο πυλώνα που θα πρέπει επίση να είναι εγγυημένο. Περιορίζομαι σε αυτέ τι παρατηρήσει. πολλά ακόμα μπορεί κανεί να πει, αλλά θα έχουμε και τη δυνατότητα στη διάρκεια τη συζήτηση να εξετάσουμε τι διάφορε επιτυχίε. Ε, well, thank you very much for... Ο πρόεδρο. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ξεκάθαρη εισήγησή σα για το σημαντικό μα θέμα. Και τώρα είναι το λόγο κυρία Χάνσλη. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ε, κυρία Χάνσλη. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να σας πω τι πρεσβεύει η κυρία Πετικάνη. Μου ζήτησε να τοποθετηθώ στη θέση της γιατί δεν μπορούσε να παραστεί. Αυτό το οποίο θέλει να σας πει αφορούν την Λευκή Βίβλο και τις συντάξεις. Ή ε, στα συμπεράσματα που αφορούν το Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέμησης της Φτώχειας και του Γενικού Αποκλεισμού ε, είχε προβλεφθεί για τους ε, ηλικιωμένους ότι εκείνοι είναι τα επικίνδυνα, ε, και εκείνοι κινδυνεύουν να πέσουν σε φτώχεια. Και γι' αυτό σας λέω, είναι πάρα πολύ βασικό πώς θα εξασφαλίσουμε κάποιες βιώσιμες και επαρκείς συντάξεις στο μέλλον. Ακριβώς βέβαια, γιατί τώρα μας έχει χτυπήσει η κρίση. Έχουμε βέβαια τώρα την σφαιρική αυτή προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οπότε θα πρέπει να δούμε πώ θα εξασφαλίσουμε τέτοιε συντάξει οι οποίε να είναι επαρκεί, οι οποίε να είναι ε, βιώσιμε. <clears throat> Επίση, ήδη ο εισηγητή μα τα είπε και κύριε Παιδικά είναι συμφωνία ει το εξή. Θα πρέπει να βελτιωθεί η διασυνοριακή συνεργασία και έτσι να μπορέσουμε να δούμε πώς θα έχουμε έχουμε αυτή την εξασφάλιση, την επιθυμητή των σύνορων παντού. Όλα είναι και περισσότεροι. Μετακινούνται πάνω από τη μία χώρα στην άλλη κατά διάρκεια αδειοδρομία του. Επομένω, <clears throat> θα πρέπει να δούμε πώ θα συνδυάσουμε τα συνταξιωτικά δικαιώματα. Επίση τώρα, όσον αφορά τι υπηκουρικέ συντάξει, όπω σήμερα έχει η κατάσταση, Αυτά τα τα ταμεία έχουν σημασία μεγάλη. Κύριε Πετικάνη θα ήθελε όμως να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Επίσης, όσον αφορά ε, παραγωγικά και υγιή γεράματα. Κυρία Πετικάινεν, έχει επεξεργαστεί αυτό το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά κάποιες εκστρατείες συνειδητοποίησης για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα συνδυάσουμε αυτού του είδους ε, την οικονομική κατάσταση με την επαγγελματική, με τον επαγγελματικό βίο, ιδίως προ την δύση τη επαγγελματική καριέρα, οπότε ακριβώ, όσον αφορά ε, την κυρία Πετικάνη θα πρέπει εδώ να βάλω τελεία, αυτά έχει να παρατηρήσει και επίση με μεγάλη μα χαρά ε, θα, θα, θα, θα τις διαβιβάσω όλα όσα είπατε και θα σας απαντήσει στην επόμενη συνάντηση. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Κύριε Χαντλίκ σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τώρα το λόγο λαμβάνει ο κύριος Μάντερς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο κύριος Κρότσμαν δεν μπόρεσε να παραστεί και συμπαθάτε τον και εγώ με χαρά μου να τον αντικαταστήσω. The, uh, directive, uh, um... We Συζητούμε για την ελόγω οδηγία μέσα σε μια συγκυρία κρίση. Και για αυτό το λόγο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το πώ θα κάνουμε πιο ευέλικτε τι συντάξει για να προωθηθούν τα αποτέλεσματα τη κρίση με τον καλύτερο τρόπο. Έχουμε 27 διαφορετικά στεσιωτικά συστήματα και φυσικά διαφορετική φορολογία και κάποια κρατημέλη έχουν μια, ένα σύστημα πολλαπλών πυλώνων και ο Σκοφράτη ήδη μας είπε ότι θα πρέπει να α, κατοχυρώσουμε κατά τον τρόπο του ηλικιωμένους από πολλές μεριές, όχι μόνο από κρατικέ συντάξεις αλλά και από ιδιωτικέ ε, και άλλου είδους ε, λύσεις μέσα από τη σταθερομία του. Γιατί σε πάρα πολλά κράτη-μέλη τώρα υπάρχει πρόβλημα πάρα πολύ μεγάλο με τις Άρα θα πρέπει εδώ πέρα κάτι να κάνουμε να στηρίξουμε το οικοδόμημα το συνταξιδοτικό μέσα στην κρίση βέβαια όλα αυτά είναι δύσκολα. Τώρα οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορούν ιστορική αγορά, οικονομία κλίμακας, αποτελεσματικότητα, πάρα πολύ θετικά όλα αυτά. Όμως στις κάτω χώρες, στην πατρίδα μου, οι περισσότερες συντάξεις προέρχονται από κάποια ταμεία τα οποία επενδύουν σε διάφορα προϊόντα τα οποία βοηθούνται από την ε, ενιαία αγορά. Προσοχή, επομένως, ότι κάνουμε να μην παραβλέψει τα οικοδομήματα που ήδη έχουν στηθεί, ήδη λειτουργούν στα κράτη-μέλη. Προσοχή, επομένως. Να δούμε τι άλλο, τι άλλο. Α, ναι όσον αφορά την ασφάλεια, την ασφάλεια των συντάξεων, θα πρέπει να προσέξουμε το τίμημα που θα καταβάλουμε, διότι δεν θα πρέπει να επιβαρύνουμε τις επιχειρήσεις, γιατί μέσα στην κρίση θα χτυπήσουμε την ανταγωνιστικότητά τους. What? Yeah, that's who should pay Somebody to pay And... Ποιο, Ποιο όμως θα πληρώσει. Ε, βέβαια κάποιος θα πληρώσει, αλλά εάν οι εταιρείε δεν είναι κερδοφόρες, ε, τι θα κάνουν. Δεν μπορούν να ε, πληρώσουν. Θα, θα, θα χρεοκοπήσουν. Ε, πώς θα βελτιωθεί η οικονομία. Ο κύριο Κρότσμαν επίσης μου είπε ότι κάτι θα πρέπει να κάνουμε όσον αφορά Τι συντάξεις. Και θα πρέπει επομένως να δούμε και μήπως βοηθούν και τα προγράμματα που θυμίζουν τις ασφάλειες ζωής και επίσης δεν προτείνεται να προχωρήσουν προς ε, λύσεις όπως το, η δεύτερη συμφωνία για την πτώχευση αλλά θα πρέπει με συγκρίσιμους κανόνες να ρυθμίσουμε και συγκρίσιμα προϊόντα. Εν κατακλείδη, Α εστιάσουμε προσοχή μα στη βελτίωση τη τουρκική αγοράς. Να δημιουργήσουμε ανάπτυξη και τότε θα μπορούμε να στηρίξουμε τις συνταξει. Άρα και η Επιτροπή μας και η γενικότερη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει αυτό να προσέξει. Και ο Σκρόιτσμαν με χαρά του να συνεργαστεί με τον εισηγητή και τους σκιώδεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Αναφέρονται τρία πράγματα εδώ πέρα. Το ότι πρέπει να δούμε τα σαλίστικα ταμεία σε ένα είδος εξασφάλισης που θα πρέπει να εκπληρώνουν τις ε, υποχρεώσεις της οδηγίας Φερικιότητα 2. Αυτό θα οδηγήσει σε χάος γιατί υπάρχουν συστήματα του δεύτερου πυλώνα που υπάρχουν σε πολλές χώρες όπου υπάρχουν πάρα πολλές ε, διασφαλίσεις και διαταραχθεί το σύστημα εάν πάμε στην ε, φερικιότητα 2. αν ε, έρθουν και σε εξασθενημένη μορφή ε, η πρόταση της Κομισιόν θα οδηγηθούμε σε τεράστια άλυψη, σε τεράστια αύξηση των απαιτούμενων κονδυλίων που θα πρέπει να ε, διακρατούνται. Αυτή τη στιγμή στην Ολλανδία παραδείγματο χάρη είναι γύρω στο 50% και θα έχουμε τεράστια αύξηση. Οπωσδήποτε βεβαίως θα πρέπει να βελτιωθεί η οδηγία όσον αφορά τους ορισμούς αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτά τα οποία ισχύουν για τι ασφαλίσει να ισχύουν και για τα συνταξιότητα κατά μία δεύτερον, το να υπάρχει μια φορητότητα των συντάξεων, νομίζω πως δεν υπήρχε πλέον ζήτημα κενών στην συνταξιοδοτική κάλυψη ε, και πως ήταν σαν να ήταν κανείς ασφαλισμένος στο ίδιο ταμείο συνεχώς. Βεβαίως μπορούν να υπάρξουν ε, βελτιώσεις ε, για τη διαφάνεια και την ε, διαδοχική όπως λέμε ασφάλιση για το πώς λειτουργεί το σύστημα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης ζητήσαμε ως Επιτροπή να ερευνηθεί ποιες είναι οι φορολογικές και οι δημοσιονομικές συνέπειες όταν κάποιος δεν πληρώνει παραδείγματο χάρη φόρο στις εισφορές αλλά όταν λαμβάνει την σύνταξη. Και η κατάσταση, διαφορεί, και η κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα. Π.χ. κάποιος μπορεί να πάει σε μια χώρα, να φύγει από μια χώρα στην οποία δεν φορολογείται η σύνταξη και να πάει σε άλλη στην οποία φορολογείται. Κάπως πρέπει να αντισταθμιστεί αυτό. Γιατί βεβαίως έχουμε συστήματα κεφαλαιοποιητικά και διάφορα, α, διαφόρων Οπότε το να ε, μεταβεί κανεί από το ένα σύστημα, από τη μία χώρα και από το ένα σύστημα στο άλλο, ε, έχει κάποιες συνέπειες και κάτι άλλο. Ο εισηγητής ανέφερε την ηλικία συνταξιοδότησης. Εμείς είπαμε πως θα πρέπει βεβαίως και στο μέλλον να είναι βιώσιμες οι συντάξεις. Ε, νομίζω καλό είναι έτσι για να μην αναφερθούμε σε τίποτα άλλο, αλλά θα πρέπει να τονίσουμε πως οι άνθρωποι θα πρέπει να μπορούν να, δουλω... να δουλεύουν μέχρι την ηλικία συνταξιοδότησης και αυτό δεν συμβαίνει. Όσα άτομα είναι πάνω από 60 δεν βρίσκουν δουλειά. Υπάρχει πρέπει να υπάρχει και υποχρέωση των ε, εργοδοτών να απασχολούν και ηλικιωμένους, πιο ηλικιωμένους εργαζόμενους για να φτάσουν στην ηλικία συνταξιοδότησης. Και όταν γίνει αυτό μπορούμε να μιλήσουμε μετά και για την ε, γύρανση του πληθυσμού. Αυτές ε, τις παρατηρήσεις έχω και εύχομαι καλή επιτυχία στον εισηγητή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λίγα λόγια και από μένα προσωπώντας τον κύριο Στράιτσεκ που είναι σκιώδης για την ομάδα μου πρώτα απ' όλα να συμφωνήσω με αυτά τα οποία είπε ο κύριος De για τα σοβαρά προβλήματα που ε, υπάρχουν με τις τωρινές συζητήσεις στην Κομισιόν για την σημαντική αύξηση απαιτήσεων χρηματοδότησης για τα υφιστάμενα συστήματα συνταξιοδότησης ε, με σταθερές εισφορές. Εάν γίνει απέτηση αυτό, θα ε, βγάλει τελείως ε, το κεφάλαιο που θα έπρεπε να επενδύεται στις εταιρείε. Νομίζω λοιπόν πως δεν έχει αποδειχθεί η ανάγκη μια τέτοια αλλαγή. Ε, Εμεί οπωσδήποτε στον Ηνωμένο Βασίλειο αυξήσαμε τι απαιτήσει για τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Αλλά πολλέ μικρομεσαίε επιχειρήσει ε, έχουν σοβαρέ ε, συνταξιοδοτικέ υποχρεώσει και επενδύουν στα συνταξιοδοτικά τα μία όσα επενδύουν και σε όλα, σε όλα τα υπόλοιπα. Και μην ξεχνάμε ότι ό,τι κερδίζει ο ένας δεν το χάνει κάποιος άλλος ή οι εισφορές αυτές με κάποιο τρόπο πρέπει να δημιουργηθούν και πρέπει να δημιουργηθούν ε, στην πραγματική οικονομία. Και πολλοί από εμά έχουμε επενδύσεις ε, σε σε συνταξιωτικά ταμεία που επανεπενδύονται στην πραγματική ε, η οικονομία επίσης. Ε, πρέπει να το δούμε λοιπόν ε, στο πλαίσιο του γενικότερου οικονομικού αντικτύπου και συνεπειών που θα έχει. Έχοντας όμως τονίσει αυτή τη συγκεκριμένη πτυχή, νομίζω πως ο αριθμός των χωρών που επηρεάζονται δεν είναι μόνο η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά νομίζω και για τη Γερμανία και άλλες χώρες επηρεάζονται. Θα ήθελα λοιπόν κάποιες περισσότερες ε, λεπτομέρειες. Υπάρχουν και κάποιες σημαντικές προτάσεις που πρέπει να στηρίξουμε εδώ πέρα, ειδικά αυτά τα οποία ανέφεραν οι συνάδελφοι ε, για το ότι ε, οι πολίτες οι οποίοι μπαίνουν στην αγορά εργασίας πρώτη φορά πρέπει να ενημερωθούν για το να κάνουν ε, μακροπρόθεσμα το κουμάντο τους. Γιατί βεβαίως η αύξηση του προσδόκιμου ζωής σημαίνει πως οι συνταξιούχοι θα έχουν συντάξεις για πολύ περισσότερα χρόνια από όσο είχε προβλεφθεί. Και βεβαίως η συνέπεια ε, είναι πως θα δουλεύουν πολύ περισσότερο. Κοιτάξτε και εγώ μόλις έγινα 65, ε, λίγο μετά την κυρία Βάιλερ. Με, με συγχωρείτε τώρα που αποκαλύπτω την ηλικία σας, αλλά έχουμε ξεπεράσει αυτό το ορόσημο και ε, μας απασχολεί πλέον το μέλλον μας και η υγιής γύρανση. Η κυρία Βάιλερ, βλέπω, θέλει να μιλήσει, Ταραμπέλα. Θέλετε να, να παραμείνετε και μετά θα επανέλθουμε στον κύριο Κομφεράτη. Ευχαριστώ. Εγώ μόλις έκλεισα τα 49, μπαίνω δηλαδή στο 50ο έτος της ηλικίας μου και αρχίζω να σκέφτομαι τη σύνταξή μου ε, με νυφαλιότητα. Να πω τις παρατηρήσεις μου. Ε, εδώ είμαστε σε μια χώρα όπου υπήρχαν περισσότερα περισσότερο ενεργητικό για τους συνταξιούχους ε, από ότι για τους ε, εργαζόμενους. Θα πρέπει λοιπόν να ξανασκεφτούμε το μηχανισμό. Τρεις παρατηρήσεις έχω να κάνω ε, σε σχέση με την εισήγηση του Σέργιο Κομφεράτη. Θέλω να επιμείνω, τα πράγμα που δεν το κάνει το Λευκό Βιβλίο, σε αυτό που κάποιοι μίλησαν για προσδόκιμο ζωής. Οι γυναίκες ζουν περισσότερο, αλλά συνήθως ε, έχουν περισσότερα προβλήματα λόγω μητρότητα, α πούμε. Αλλά ε, το προσδόκιμο ζωή δεν είναι το ίδιο για όλα τα επαγγέλματα. Ένα καθηγητή πανεπιστημίου συνήθω θα ζήσει περισσότερο από ότι ένα ανθρακορίχο ή ένα εργάτη στη βαριά βιομηχανία. Τώρα, βέβαια, η σταδιοδρομία 40-45 ετών ε, στην ίδια δουλειά είναι σπάνια. Θα διακρίνουμε διάφορα κομμάτια σταδιοδρομία που γίνονται σε πολύ δύσκολα επαγγέλματα, βαριά επαγγέλματα. Ε, να επιβεβαιώσω τη δεύτερη λοιπόν παρατήρησή μου τώρα ότι, που σχετίζεται με το ποσοστό απασχόλησης. Το ποσοστό απασχόλησης ας πούμε για το κομμάτι το ηλικιακό κοντά στη συνταξή, δηλαδή 55 μεταξύ 5 ετών διαφέρει. Στην Βέλγιο, πούμε, δουλεύουν το λιγότερο οι άνθρωποι ανάμεσα στα 55 και τα 65. Το ποσοστό απασχόλησης είναι μόλις 36%. 36% των 55 με 65 εργάζονται στο Βέλγιο. Και αυτό δεν οφείλεται μόνο στις βιομηχανίες που αναδιερθώνονται και υπάρχει και το θέμα των απολύσεων σε διάφορα βιομηχανικά ε, έργα, ε, μέρη είναι και το θέμα των ασφαλίσεων. Θέλουν να τους ενθαρρύνουν να φεύγουν για να παίρνουν τους νέους, τους οποίους πληρώνουν πολύ λιγότερο. Και αντί να αυξήσουμε λοιπόν, αυξήσουμε, λοιπόν το, ε, την ηλικία συνταξιδότησης, να, κάνουμε, να βάλουμε στη δουλειά ένα σωρό κόσμο που μπορεί να δουλέψει ακόμα και που βγήκε πολύ νωρίς στη σύνταξη υποχρεωτικά. Και τρίτο σημείο είναι η βιωσιμότητα να εγγυηθούμε ένα σύστημα σίγουρο. Δεν το γνωρίζω πολύ καλά το σύστημα το συνταξιδοτικό, αλλά είχα διαβάσει ένα έργο, ένα ε, άρθρο όταν ε, εκείνο το πετρελοφόρο άρχισε να μολύνει τις αμερικανικές ακτές ε, λόγω του ναυαγίου τα νούμερα για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος θα κόστιζαν δισεκατομμύρια. Όμως το ίδιο πρέπει να σκεφτούμε με τη σύνταξη. Ας πούμε αυτά ε, ισχύει Ας πούμε για το βρετανικό σύστημα συντάξεων δεν μπορεί ένα ναυάγιο να θέτει σε κίνδυνο ολόκληρο το συνταξιδοτικό σύστημα των Βρετανών ναυτικών. Εντάξει να είναι στην, ε, στο χρηματιστήριο, αλλά θα πρέπει να υπάρχει εξασφαλισμένη σύνταξη τη στιγμή που ο εργαζόμενος βγαίνει στη σύνταξη. Ευχαριστώ. Βάιλερ. Ε, είμαι σύντομη. Θα περιοριστώ. Το εξή. Εκεί όπου θεωρώ πως έχουμε υποχρεώσεις για να δράσουμε. Παραδείγματο χάρη, όπω είπε ο κύριο Ταραμπέλα, όταν συνταξιοδοτικά ταμεία επηρεάζονται από διασυνοριακά γεγονότα, πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να, να δώσει κάποιες εγγυήσει. Αλλά, εάν δεν μιλάμε για διασυνοριακές πτυχές και την κινητικότητα των εργαζομένων, πρέπει να είμαστε κάπως επιφυλακτικοί. Εμένα δεν με ενθουσιάζει πως, δεν θέλω να πω υπαγορεύει, αλλά συνιστά επιμόνως σε κράτη-μέλη κομισιών να αυξήσουν τη ηλικία συνταξιοδότηση δεν μου αρέσει καθόλου. Όλα τα κράτη-μέλη ξέρουν πόσο ακαθόδες είναι αυτό το θέμα και οι εθνικοί βουλευτές δίνουν αγώνα για να βρουν μια ισορροπία μεταξύ του υψηλότερου κόστους και του αυξημένου προσδόκιμου ζωής. Και ε, τώρα από τις Βρυξέλλες να έρχεται η διαταγή ας πούμε, κάνα αυτό ή το άλλο, δεν είναι σωστό. Με εξαίρεση, όπως είπα, τις διασυνοριακές πτυχές που πρέπει να προστατεύσουμε τον καταναλωτή. Είμαι δε πεπισμένη πως οι εθνικοί βουλευτές ε, έχουν συνέστηση της ευθύνης ε, ή τουλάχιστον της δικής μου ομάδας ε, το, της ευθύνης του να μην είναι φτωχοί οι ηλικιωμένοι. Αυτό όμως είναι αποστολή των Εθνικών Κοινοβουλίων και πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί αν δούμε το τι λέγεται και στο γαλλικό προεκλογικό αγώνα του χρόνου έχουμε και στη Γερμανία εκλογές. Βλέπω το τι ε, συζητήθηκε στην Ελλάδα. Οπωσδήποτε πρέπει να αλλάξει κάτι, αλλά αυτό πρέπει να το κάνουν οι Έλληνες ε, μόνοι τους. Δεν είναι σωστό εμείς να υπαγορεύουμε ε, και μέσος ακόμα πόσο ψηλή ή χαμηλή θα είναι η ηλικία συνταξιοδότησης. Υπάρχει Ιωσή Τσέγγεν εδώ πέρα από την Γενική Διευθύνση Απασχόληση, αλλά φοβάμαι πω δεν έχουμε χρόνο. Όταν παρουσιάστηκε με τον κύριο Κοφεράτη θα το συζητήσουμε. Κύριε Κοφεράτη, λοιπόν, θέλετε να, να ολοκληρώσετε και μετά θα δούμε και το χρονοδιάγραμμα τη εκθεσή σα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα κάνω σύντομες παρατηρήσεις να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις υποδείξεις που μου έκαναν και που θα τις χρησιμοποιήσω στην σύνταξη της πρότασης. Ε, προτείνεται ε, και εκ νέου, όχι τυχαία, το ε, θέμα της σταθερότητας των συνταξιδοτικών ε, συστημάτων, των συστημάτων πρόνοιας σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ελπίζω να ζούμε ακόμη περισσότερο, όμως η αύξηση του προσδόκιμου ζωής δεν πρέπει να επιφέρει κινδύνους για το σύστημα προνοίας. Αν θέλουμε να εγγυηθούμε στον κόσμο μια κατάλληλη σύνταξη και όχι μια... Δήθεν σύνταξη. Γιατί τα προβλήματα τα οποία εντοπίστηκαν ε, επιβεβαιώνουν ότι το να έχει κανείς μια σύνταξη είναι πολύ σημαντικό ε, για εκατομμύρια κόσμο. Οι δρόμοι που έχουμε να διαλέξουμε είναι δύο, δεν είναι 100 όσον αφορά την κοινωνική πρόνοια. Δηλαδή, σταδιακή αύξηση της, της, ε, του ορίου δεξιδότησης ξέρουμε και ευτυχώς ε, οι συνθήκες ζωής είναι καλύτερες από για τους γονείς μας ας πούμε και ε, από την άλλη πλευρά να αλλάξουμε τα συστήματα κατανομής. Τα συστήματα κατανομής όμως οδηγούν σε χαμηλότερες αξίες. Κατά συνέπεια, και είναι η δεύτερη πτυχή, είναι απαραίτητη, απαραίτητος ο δεύτερος πυλώνας από την αρχή που, της ζωής του κάθε ανθρώπου. Με ειδική πρόνοια βέβαια και πρόβλεψη για τις γυναίκες. Ε, ε, όσον αφορά όμως το δεύτερο πυλώνα, το βασικό θέμα για μας, για την Επιτροπή μας, είναι να λύσουμε ή να δώσουμε κάποιες ενδείξεις για την επίλυση το θέμα τους που αφορά τη δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων. το Πρόβλημα προκύπτει λόγω της δυνατότητας ελεύθερης κυκλοφορίας των ατόμων ώστε αυτή η αναγκαστική ε, ε, ε, εξοικονόμηση γιατί είναι χρήματα που δίνουν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες να μην εκτίθεται στους κινδύνους του οικονομικού κύκλου. Θα πρέπει λοιπόν να δίνονται εγγυήσει στους ανθρώπους, στα άτομα και αυτά είναι συγκεκριμένες ε, φορολογικές παρεμβάσεις και επενδύσεις όχι κερδοσκοπικές αλλά σταθερές και διορθωτικές, τόσο ώστε κανένας, κανένας ξαφνικά ε, να μην εξαφανίζεται, να μην εξαφανίζονται τα λεφτά γιατί ήταν ε, ε η διαχείριση των ταμείων. Ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ και περιμένουμε πώς και πώς να δούμε το κείμενό σας. 3 Μαΐου, 13 Μαΐου παρουσίαση, 12 Ιουνίου είναι η για της τροπολογίας και στις 10 Ιουλίου θα γίνει η ψήφιση. Περιμένουμε να δούμε. Ο κ. Λίχτεμπεργκ είναι εδώ από την ε, αρμόδια Γενική Διεύθυνση, αλλά δεν είχαμε το χρόνο να τον ακούσουμε και εκείνο. Ακούσαμε πάρα πολύ. Και τώρα. Πάμε στην εκθέση Μπουσούτιλ. Σχέδιο κειμένου. Καλώ Ξέρω ότι έχετε υποχρεώσει και σε άλλε επιτροπέ. Και πάρα πολύ τα πήγαμε. Είπα να συζητήσω το θέμα σα τώρα που φτάσατε. We've had some useful amendments from Έχουμε και σχέσει τροπολογία τη εκθεσή σα. Σάντσες Φανχόβεν είναι η εκπρόσωπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με μεγάλη μας χαρά να σας δώσουμε το λόγο. Έχουμε εδώ όλους τους ισχυροσυγητές, από εδώ είναι παρόν ο κύριος Μπίλαν, οι υπόλοιποι δεν είναι εδώ, τόσο να τα συζητήσουμε. Έχετε το λόγο κύριε Συγητά. Μπουσούτε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η έκθεση που συνέταξα σε σχέση με τις επιδόσεις της εσωτερικής αγοράς φτιάχτηκε σε συνέχεια της 22ης ε, αντίστοιχης έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και από τότε, όπως είπαμε και την τελευταία φορά, όταν ανταλλάξαμε απόψεις, είχαμε κάποιες ε, αλλαγές και από τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε την 23η έκθεση και το ετήσιο check-up. Έχουμε πει στην 10η έκθεση όσον αφορά και τα προβλήματα της τελικής αγοράς. Οπότε, επιτρέψατε μου να σας ε, πω δύο λόγια σε σχέση με τις 66 αυτές προπολογίες ε, που έχουν υποβληθεί για την έκθεσή μου. Οι περισσότερες εξ αυτών με τον πίνακα αποτελεσμάτων αφορά την ε, ενημέρωση, επικαιροποίηση για να καλύψουμε τις ε, εξελίξεις που σας προανέφερα. Οπότε τα πράγματα είναι αρκετά απλά, δεν έχουμε εδώ κάποια σημεία επίμαχα, οπότε θα πρέπει να σας αναφέρω ότι περισσότερες από τις τροπολογίες πάνε προς την ίδια κατεύθυνση, οπότε Όλες, όλες μπορούμε να τις καλύψουμε. Και τις 66. Πάρα πολύ σωστό αυτό. Να ανέβει εδώ πέρα ειρήνη, γαλήνη, τέλος πάντων. Μέσω αυτών των τροπολογιών επίσης είχαμε και την ευκαιρία να δούμε τι άλλα λέει σε, αυτή, σε αυτό το, το, το, το την ετήσια ε, έκθεση Ευρωπαϊκή Επιτροπής για την ε, διακυβέρνηση και συγχαρητήρια για την έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μένα είναι ανταπόκριση σε αυτά τα οποία θέλουμε, ούτως ώστε να συνδυάσουμε ε, ό,τι έχουμε από εδώ και από εκεί και να έχουμε καλύτερο συνενισμό. Και έτσι μπορούμε να καλύψουμε ό,τι θέλουμε. Επομένω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να δημοσιεύσει χωριστές εκθέσει για διαφορετικά στοιχεία τα οποία περιέχεται σε αυτή την ετήσια εκθεσή της σε αυτό το σε αυτό πίνακα αποτελεσμάτων και κατά αυτόν τον τρόπο να έχουμε τακτές εκθέσεις και να είναι αναδιατήρια, όχι αυτές οι εκθέσεις δημοσίευσης και έτσι να έχουμε μια σφαιρική, συντονισμένη προσέγγιση και να μην γυρίσουμε προς ε, κατάτμιση των ιδιών μας. Οπότε, Σα το επισημαίνω αυτό να το προσέξουμε. Επίση, θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει περισσότερο, τόσο ώστε να δώσει στον κόσμο ένα ολοκληρωμένο πακέτο δέσμη μέτρων όσον αφορά ε, μια προσέγγιση που θα βοηθήσει να επιληθούν τα προβλήματα που αφορούν την εσωτερική αγορά. Όντω, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδο στο παρελθόν στο πρόσφατο παρελθόν και ιδίω όσον αφορά αυτή την μονοπευθυντική θηρίδα. Είχαμε την οδηγία για τις υπηρεσίες. Solvit και Europe Direct αυτές, αυτά τα κείμενα και πρόκειται τελικά αυτή η οδηγία για τη φερικαιότητα ε, και άλλοι για τις υπηρεσίες τελικά είναι διόψη του ίδιου νομίσματος να δούμε τι και πότε θα χρησιμοποιούν οι Ευρωπαίοι. Άρα θα πρέπει να σταματήσει να υπάρχει η σύγχυση και θα πρέπει να μην πηγαίνει κανείς στο λάθος, στη λάθος πηγή ή επίσης θα πρέπει να πηγαίνει κάπου που τελικά να το προσφέρει τη λύση. Οπότε θεωρώ ότι πρόκειται για έναν φραγμό στο έργο τη συμπορία τη ειδικής αγορά. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να το καταπολύουμε αυτό το, το, αυτό το, το, το, το εμπόδιο. Και οι τρόπολογίε βοηθούν. Οπότε και θα πρέπει να δοκιθούμε σε καλύτερη συνεργασία μεταξύ των επιμέρους υπηρεσιών. Επίσης, να δούμε τι αποδίδει καλύτερα, ιδίω όσον αφορά την ε, έκθεση που προανέφερα γιατί μια άλλη όψη του νομισματος είναι, όπως το βλέπω εγώ, το ότι ακόμη οι Ευρωπαίοι δεν ξέρουν τι να κάνουν. Όταν να αντιμετωπίσουν το σε ποιον πρέπει να απευθυνθούν όταν θέλουν να επιληφθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά και δεν είναι το πλήρω εξωτερικό είναι η υπηρεσία για την εσωτερική αγορά. Αλλά όμω ακόμα, ακόμα δεν ξέρουν τι να κάνουν όταν είναι η ώρα του να απευθυνθούν στην Ευρώπη. Επομένω, πρόκειται για πρόβλημα το οποίο πηγάζει από το ότι ακόμα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη γραφειοκρατία, ούτω ώστε οι πολίτε δεν ξέρουν να κάνουν τώρα. Καμιά φορά πρέπει κανεί να ζήσει με το πρόβλημα, να το ανεχθεί και όχι να προσπαθεί να το λύσει και έτσι να παρακάμψει το λαβύρινθο των διαφορετικών υπηρεσιών. Αυτή είναι η υπόψή μου. Αλλά το λένε και οι τροπολογίε συνάδελφοι. Είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση. Θα πρέπει επομένω να αυξήσουμε την προσβασιμότητα και θα πρέπει επίση να υπάρχει άμεση επαφή με κάποιου ε, υπηρεσίε που όντω μπορούν να βοηθήσουν τον κόσμο. Και έτσι να άρουμε τα, τα, τα εμπόδια για την ιστορική αγορά. Αυτά. Βεβαίω και εδώ πέρα έχουμε πάρα πολλέ δυνατότητε. Και φυσικά ε, δεν εξαντλείω ε, τα θέματα η εκκλησία μου. Προσπαθούμε πάντως να δούμε τι μπορούμε να βρούμε. Οπότε παρακαλούμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όποτε μπορεί, ας επανελθεί για να δούμε πώς μπορεί να λυθούν αυτά τα προβλήματά μας και έτσι να έχουμε μία ισχυρή εσωτερική αγορά. Αυτά όσον αφορά τις 66 τροπολογίες που έλαβα. Να ευχαριστήσω επίσης και τους συναδέλφους για τη συνεργασία τους γιατί νομίζω ότι έχουμε εδώ πάρα πολύ σημαντικές ε, συνεργατικές προσπάθειες ε, προς μία ε, λύση στην Επιτροπή μας. Και σε αμέσως μερες μέρες θα κατεβάσουν προτάσεις για τις συμμετοχές των του τουλάχιστον πέντε. Και έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε κάποιες πιο συνεκτικές τροπολογίε. Εδώ θα βάλω τελεία και θα περιμένω να ακούσω την αντίδραση των συναδελφών. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρος. Οπωσδήποτε συμφωνώ μαζί σα για την κατεύθυνση των πραγμάτων. Ευχαριστώ και τους κοιόδης συγητές για την ενημέρωση τη έκθεσης που είναι πάντα το δύσκολο την επικαιροποίηση της έκθεσης, οπότε ας δούμε τι έχουν να πούν οι σκιώδεις εισηγητές. Ας ξεκινήσουμε με τον Κορέα πως Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπουσούτιλ για την παρουσίασή του και χαίρομαι για το ότι είναι ανοιχτός σε ε, τροπολογίες από τους ηγητές και άλλους έχουμε 66 τροπολογίες που πηγαίνουν λίγο πολύ στην ίδια κατεύθυνση Προσπαθούμε λοιπόν να δούμε ότι γίνεται όσον αφορά τη μεταφορά και σε ταχύτητα και σε ποιότητα για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η ανακοίνωση για τις κυβερνήσεις και την εσωτερική αγορά του 2011, μας δίνει μια χρήσιμη γενική εικόνα της εσωτερικής αγοράς. Μας δίνει μια γενική εικόνα του σε ποιο βαθμό πηγαίνουμε σε μια πλήρη ε, λειτουργικότητα και βεβαίω αυτό είναι ένα χρήσιμο έγγραφο για την λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Έχουμε διάφορα μέσα στη διάθεσή μας όπως το Solvit ε, και άλλα μέσα για να υπάρχουν ε, πληροφορίες στην διάθεση των πολιτών για την καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα κάποιας αδράνειας στα κράτη-μέλη όσον αφορά την μεταφορά των οδηγιών. Εδώ πέρα νομίζω πως χρειάζεται καλύτερος έλεγχος ε, από τις Βρυξέλλες για το, τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Η Επιτροπή μας θα πρέπει οπωσδήποτε και η Κομισιόν και το Συμβούλιο να δείξει πως ε, είναι υπέρ της σωστής εφαρμογής ε, της ε, εσωτερικής αγοράς. Um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Λόκεγκαρτ. Να συγχαρώ τον συγητή πρώτα απ' όλα. Οι 66 τροπολογίες δείχνουν πως ήταν σωστή η απόφαση να αναβληθεί η έκθεση για να έχουμε και τις τελευταίες εξελίξεις στον πίνακα βαθμολογίας αλλά και μια γενική εικόνα των εξελίξεων. Νομίζω πως οι τροπολογίες το δείχνουν αυτό. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Αν μου επιτρέπετε, είναι λυπηρό το ότι άλλαξε προθεσμία υποβολής τροπολογιών και δεν πρόλαβα να υποβάλω τροπολογίες. Ε, φταίω και εγώ βεβαίω. αλλά ίσω στο μέλλον θα μπορούσαμε να έχουμε μια καλύτερη ενημέρωση. Ε, να πω λίγα λόγια για το τι σκόπευα να καταθέσω. Θα πρέπει να τονίσουμε πως η αρχή του να κατονομάζουμε θα πρέπει να αναφερθεί ρητά το κατόφλι εφαρμογή του 1% θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα εφαρμόζουν όλα τα κράτη-μέλη και να το χαμηλώσουμε νομίζω στο μισό της εκατό. Η προσέγγιση αυτή του να κατανομάζουμε είναι ένα ισχυρό εργαλείο, πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη. Το ίδιο ισχύει και όταν μιλάμε για την μείωση ε, της ε, καθυστέρησης μεταφοράς. Ελπίζω λοιπόν ο εισηγητής και οι να αποδεχθούν κάποιες από αυτές τις ιδέες. Αυτά και ευχαριστώ πάρα πολύ. Okay, well, thank you. I, I wasn't aware of the problems you talked about, but I'm sure that... Τα γνωρίζω αυτά τα οποία είπατε. Είμαι σίγουρος πως ο κύριος Μπουσούτιλ ε, θα λάβει υπόψη τις τροπολογίες σας. Θα είμαι σύντομη, ευχαριστώ τον συγητή, ευχαριστώ και για τις ε, τροπολογίες. Είναι πολύ καλές. Βεβαίως ο χρόνος πιέζει. Οπότε θα ε, τελειώσω το πέρα την παρέμβασή μου. Ευχαριστώ κύριε Σπίλα. Ευχαριστώ. θα είμαι και εγώ πάρα πολύ σύντομος. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική αυτή έκθεση. Έχω καταθέσει 15 τροπολογίες. Ε, η πολιτική μου ομάδα στηρίζει πλήρως την έκθεση αυτή και αναζητούμε συμβιβασμό. Κάποιος άλλος θέλει να παρέμβει. Η Κομισιόν. Ναι. Κύριε, ο κύριος Μπουζουτήλ, λοιπόν, για να συνοψίσει και να μας πει τι θα γίνει από εδώ και μπρος. Ε, για να πάμε στην 25η Απριλίου και την υιοθέτηση. Target for adoption is for the 25th April, as you said, Mr. Chair. Ακριβώς ο στόχος, όπως είπατε, κύριε Πρόεδρε, είναι 25η Απριλίου. Πριν από αυτή την ημερομηνία, ελπίζω να καταθέσω κάποιες συμβιβαστικές ε, τροπολογίες. Ήδη βλέπω τουλάχιστον πέντε που θα προσπαθήσω να συγκεράσω διάφορα στοιχεία που υπήρχαν στις ε, τροπολογίες. Δεν μπορώ να διαφωνήσω με σχεδόν οτιδήποτε. Ε, σημείωσα αυτό το οποίο είπατε και θα φροντίσω να ε, τα βάλω σε συμβαστικές τροπολογίες. και ε, δεν, θα υπάρχει δυσκολία. Ε, με συγχωρείτε που επηρεαστήκατε από τις προθεσμίες, δεν το ήξερα, δεν το ήξερα. Οπωσδήποτε θα φροντίσω να λάβει υπόψη αυτά τα οποία είπατε στο πλαίσιο του συμβασμού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που συνεργάστηκαν έξοχα ε, για να γίνει καλύτερη η έκθεση. Ευχαριστώ. Okay, well... Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να επιβεβαιώσω πως θα ψηφίσουμε 25 Απριλίου και ε, πάμε, ελπίζουμε, στην ονομέλεια τον Μάιο. Ε, τελειώσαμε και είμαστε λίγο μπροστά από το χρονοδιάγραμμα, αλλά βλέπω πως και οι δύο εισηγητές είναι εδώ πέρα. Βλέπω και θέση ο κύριο Στανόη, ο οποίο. Ήρθε ο κύριο ο οποίο είναι παλιό φίλο και παλιό συνεργάτη του έργου τη Επιτροπή μα. Οπότε αν δεν έχετε καμία αντίρρηση, να προχωρήσουμε να πάμε στο επόμενο θέμα. Έχουμε εδώ του δύο συγκεκριτές. Κοινό Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Πολίσεων. Ο κ. Κότσμαν δεν είναι εδώ. Δεν ξέρω ποιος είναι ο σκιώδης για τους ε, πρασίνους. Η κυρία Ρούλερ θα μιλήσει. Ο κύριος Φόξ είναι ο εισηγητής ε, για το ECR. Θα, θα αντικατασταθεί. Ούτε ο κύριος Τεντεφλίδης παρίσταται. Οπότε, πρόκειται για την πρώτη επίσημη συνάντηση. Οπότε που αποφασίσαμε να έχουμε συνεισηγητές, ακριβώς όπως ε, είπαμε και για την νομική επιτροπή. Έχουμε συμφωνήσει τώρα, όπω και στην νομική επιτροπή. Έχουμε συμφωνήσει όσον αφορά τι αρμοδιότητε της μια επιτροπή και τη άλλη. Συμφωνήσαμε ποιε είναι οι αποκλειστικέ και ποιε είναι οι κοινέ αρμοδιότητε. Νομίζω τα ξέρουν αυτά οι συγκητέ. Το θέμα επομένω προχωρεί. Τώρα, κύριε Σόλμαγερ, θέλετε το λόγο, εσείς πρώτος, ή η κυρία Γκέμχαρτ, ο κύριος Μάγερ. Κύριε Πρόεδρε, εγώ είμαι Μέλο συντηρητικού κόμματο οπότε οι κυρίε προηγούνται. <laughs> Κυρία Γκέπχαρτ. Ε, δεν θα αρχίσουμε τώρα ποιο θα αρχίσει και ποιο θα, ακολουθήσει. Τέλος πάντων είμαι και υπέρ τη ισότητα. Ε, υπάρχουν και άλλα κριτήρια λοιπόν. εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκαθαρίσω το εξή. Ε, λυπούμε για το ότι δεν έχουμε την κυρία αρμοδιότητα για το θέμα αυτό, γιατί πρόκειται πράγματι για προστασία των καταναλωτών. Θα το ξαναπώ, το είπα και την προηγούμενη φορά, θέλω να το επαναλάβω ε, και σήμερα και λυπούμε ιδιαίτερα ε, για το ότι στο άρθρο 3 υπάρχει ε, αποκλειστική ευθύνη της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. Θέλω εδώ να υπενθυμίσω πως ε, εγώ έλεγα στην ομάδα μου μέχρι τέλους πως δεν συμφωνώ. Γιατί το, άρθρο αυτό εξαρτάται η διαμόρφωση ολόκληρου του κειμένου και σε τομείς ε, που είναι πράγματι προστασία των καταναλωτών. Πρέπει να γίνει ακόμα αυτή η συζήτηση στο Κοινοβούλιο και δεν έχει γίνει σωστά για το, αυτό, το 28ο καθεστώς. Το θέμε ή όχι. Αυτό είναι το θεμελιώδες ερώτημα που τίθεται. Εάν δεν απαντήσουμε όμως και δεν μπορούμε να απαντήσουμε εμείς αυτό το ερώτημα, τι να πούμε επί της ουσίας. Δύσκολα να μιλήσουμε για αυτή την έκθεση. Και να πω πως εγώ προσωπικά ως συνεισηγήτρια, δε, χωρίς να έχω συζητήσει με τον κύριο Μάιερ, θα προτιμούσα πάρα πολύ να έχουμε ελάχιστη εναρμόνιση, μια τέτοια οδηγία, αντί για ένα 28 28ο καθεστώς. Και θα ήθελα να αιτιολογηθεί εδώ πέρα. Ε, βεβαίως αυτό είναι η προσωπική μου θέση χωρίς να θέλω να προκαταλάβω την άποψη της ε, μου συνολικά. Αλλά ε, το ξέρει η ομάδα εργασία, δεν το έχουμε συζητήσει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι λοιπόν πολύ προβληματικό αυτό το προαιρετικό σύστημα γιατί είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό το οποίο θέλαμε, δηλαδή σαφήνεια για τους ε, καταναλωτές. Εγώ δεν βλέπω κάποιο πλέον έκτημα για τους καταναλωτές ε, όταν αγοράζουν κάτι ε, και ξαφνικά έχουν μπροστά τους δύο συμβάσεις και τους λένε επιλέξτε με ποιο καθεστώς θα κάνετε την αγορά. Δεν μπορώ να φανταστώ πως θα σχοληθεί κανείς ε, καταναλωτής να συγκρίνει δύο νομικά κείμενα και να πει ε, ποιο συμφέρει. Και βεβαίως η συμβουλή του εμπόρου θα είναι προς ε, το καθιστός το οποίο συμφέρει εκείνον και όχι οπωσδήποτε τον καταναλωτή. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο είμαι πολύ επιφυλακτική για το 28ο ε, καθεστώς είναι πως είναι τελείως ε, ε, θολή η σχέση του με τον κανονισμό της Ρώμης ένα όπου βεβαίως εκεί πέρα αναφέρεται πως έχει ισχύει το δίκαιο του κράτους ε, του αγοραστή. Ε, τι θα γίνει εδώ πέρα τη στιγμή που ισχύει ακόμα ο κανονισμός Ρώμη 1. Γι' αυτό, επαναλαμβάνω, και λυπούμε για το ότι το άρθρο 3 που ακριβώς αυτό το ζήτημα αντιμετωπίζει, ποια βάση έχουμε δηλαδή για το κείμενο, δεν μας λέει τίποτα. Και επίσης καθιστά λίγο πολύ παροχημένη την ενισχυμένη ε, συνεργασία και πρέπει να τα συζητήσουμε με τον κύριο Μάιερ τι θα κάνουμε εδώ πέρα για να κάνουμε ό,τι μπορούμε από την υφιστάμενη κατάσταση γιατί πρέπει να ψηφίσουμε πριν από την ε, ψηφοφορία στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων πριν ε, ρυθμιστεί αυτό το θέμα κατόπιν. Αυτά τα προβλήματα έχουμε και μας δυσκολεύουν. Τώρα, να περάσω στην, ε, στην ουσία πολύ χοντρικά ε, γιατί είναι η πρώτη συζήτηση και πρέπει να διαβάσω και το κείμενο πριν ε, τοποθετηθώ. Αλλά αναρωτιέμαι πώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα βολευτούν εδώ πέρα. Μα δεν μπορώ να συζητήσω. Δεν μπορώ να συζητήσω χωρίς το άρθρο 3. Γιατί όλα από εκεί ξεκινάνε και καταλήγουν. Είναι αδύνατον. Μα ε, τέλος πάντων, λέει εδώ πέρα πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, θα ωφεληθούν ε, εάν έχουν ένα προαιρετικό σύστημα. Αλλά λυπούμε, πως εγώ δεν το, λυπούμε για το ότι πρέπει να πω πως εγώ δεν το βλέπω αυτό. θα ε, χρειάζονται μικρομεσαίες ε, και οι μεγάλες επιχείρησεις. Μια νομική ασφάλεια, μια απλή κατάσταση την οποία θα ξέρουν. Το λένε όλες, μεγάλες μικρές επιχειρήσεις. Εμείς θέλουμε ένα απλό κείμενο και όχι πέρα δόθε και να μην ξέρουμε τι, τι μας γίνεται. Και νομίζω πως είναι επίσης λάθος να πούμε πως ε, οι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν συνεχώς 28 καθεστώτα. Εγώ μίλησα με εμπόρους που κάνουν δύο συνοριακές πωλήσει. Και μου λένε, «Ε, ξέρετε, εμείς το κάνουμε κατά περίπτωση. Καταρχήν δεν εμπορευόμαστε και με τις υπόλοιπες 26 χώρες. Κάνουμε το ένα μετά το άλλο. Ξεκινάμε από τις σημαντικότερες για εμάς χώρες και βλέποντας και κάνοντας. Αλλά να επανέλθουμε στη, στην προστασία των καταναλωτών. Να καταπιώ το θυμό μου και να σας πω τι θα κάνουμε εδώ πέρα. Η Ευρωπαϊκή Κομισιόν ε, ισχυρίζεται πως ε, στην πρόταση αυτή ε, προβλέπεται πολύ υψηλό επίπεδο δικαίου των ε, συμβάσεων. Ε, τα μηνύματα που μου ήρθαν εμένα από τα κράτη-μέλη, από κυβερνήσεις, ε, από οργανώσεις καταναλωτών και επιχειρήσεις πηγαίνουν προς την κατεύθυνση πως σε πολλά σημεία δεν ισχύει αυτό το οποίο ισχυρίζεται η Κομισιόν και πρέπει να δούμε τα θέματα αυτά. Εάν πρέπει να υποθέσω πως σε αυτά εδώ τα ζητήματα θα έχουμε ένα επιπλέον προαιρετικό σύστημα. Πρέπει να δούμε ακόμη μία φορά τα διαφορετικά επίπεδα προστασίας για να δούμε ποιες αλλαγές ε, μπορούν να γίνουν. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ. Δεν μπορώ να πω κάποια οριστικά πράγματα γιατί πρέπει να ερευνήσω. Ποια είναι τα διάφορα σημεία. Είναι πολύ πολύπλοκο το κείμενο. Και όπως συχνά στα κείμενα της Κομισιόν έχει διάφορες παραπομπές, παραρτήματα και πρέπει να το διαβάσω με προσοχή για να δω τι γίνεται ακριβώς. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Μάιερ, ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη συζήτηση που έχουμε κάνει πολλές φορές και είμαι σίγουρη πως θα συνεργαστούμε στενά και θα βρούμε μια διαδικασία, έναν τρόπο συνεργασίας θα δούμε ποιες είναι οι κοινέ μας θέσεις για να έχουμε ε, ένα σχέδιο έκθεσης και μετά θα δούμε που δεν συμφωνούμε και μετά θα κατατεθούν οι τροπολογίες äh, για να έχουμε μία βάση συζήτησης. Θεωρώ λοιπόν πως είναι ένας λογικός τρόπος εργασίας αυτός έτσι ώστε εκ των προτέρων να μπορέσουμε να καλύψουμε αρκετά πράγματα αλλά παρόλα αυτά βεβαίως θα είναι σαφές το που διαφέρουν οι ομάδες. Αυτό είναι θετικό για τους πολίτες για να ξέρουν ε, ποιες είναι οι διαφορετικές πολιτικές απόψεις. Ελπίζω να μην είναι πάρα πολλές. Είχα την εντύπωση πως ε, ε, πολιτικά είμαστε πάρα πολύ κοντά και χαίρομαι ιδιαίτερα για τον τρόπο αυτό της συνεργασίας. Είναι η πρώτη φορά που είχα τη δυνατότητα να είμαι συν εισηγήτρια. Είναι καινούριο αυτό για μένα. Και είναι μια θετική εμπειρία και σας ευχαριστώ. I think, ευχαριστούμε. Τι να σα πω, να σα πω, δεν ξέρω συμφωνώ με εσά. Εγώ πάντω πρέπει να είμαι ουδέτερο τώρα για να δούμε. Δουλεύουμε θεωρώντα ότι είναι μη υποχρεωτική αυτή η ρύθμιση. Εάν βεβαίω πέρασε από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τώρα βέβαια θα μπορούσε η κοινωνική Επιτροπή να τα ανατρέψει όλα. Τότε θα πρέπει να ξαναδιαπραγματευτούμε. Εγώ θεωρώ πάντω ότι θα συνεχίσουμε εργαζόμεθα ότι πρόκειται περί μη υποχρεωτικής ρύθμισης. There are a number of other others who question the added value of that, and I should have drawn your attention, by the way, to the fact. Αυτό ήθελα να σας επισημάνω. Επίσης, σας επισημάνω ότι έχουμε τέσσερις αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις του Εθνικών Κοινοβουλίων σε σχέση με το ότι η παρούσα πρόταση, η, αυτό το κοινό Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Πολίσεων, δεν συμβαδίζει με την επικουρικότητα. Έχουν βέβαια και τόσα άλλα για κοινοβούλια που δεν ξέρουν θέλουν να πούν. Πάντως τα σχόλια αυτά το έχετε λάβει ως κείμενα ή στους φακελός σα Και τώρα, ο συνεισηγητής, κύριος Μάγερ. Ευχαριστώ. Οι ανώτεροι μας εν τη σοφία τους αποφάσισαν να είμαστε συνεισήγητες. Εγώ το γνωρίζω από την ε, ΑΚΕ. Εκεί πάντα είχαμε συμπροέδρους, ε, συνεισηγητές. Τα προβλήματα είναι τα ίδια. Βεβαίω ε, δεν είναι τόσο απλό να καταλήξουμε πάντα σε μια κοινή έκθεση και η Εύελιν έχει δίκιο σε πάρα πολλά θέματα αρχής ε, προστασίας των καταναλωτών ε, συμφωνούμε παρόλα αυτά. Θεωρώ πως πρέπει να έχουμε ως αφετηρία πως θα είναι ένα προαιρετικό μέσο γιατί βεβαίως ε, είναι ξεκάθαρο το λέει και ο κανονισμός πως το αστικό δίκαιο είναι η υπόθεση της Επιτροπής, Δικαίων, ε, της Επιτροπής Δικαίου νομικών υποθέσεων. Οπότε πράγματι μπορούμε εδώ πέρα να συνεισφέρουμε την άποψή μας. Οπότε όπως είπαμε είμαστε συνεισηγητές, εκεί που δεν συμφωνούμε θα καταθέσουμε τις ανάλογες τροπολογίες ε, και η Επιτροπή πάλι θα προσφέρει την σοφία της και μετά η Επιτροπή ε, Νομικών Υποθέσεων θα είναι η σοφότερη από όλες και θα έχει την τελική, τον τελικό λόγο. Θεωρώ πως, ε, για να πω και κάποια πράγματα, πως το προαιρετικό μέσο είναι καλύτερο από την ελάχιστη εναρμόνιση. Η Γερμανία είναι μία από τις τέσσερις χώρες που ανέφερε ο πρόεδρος ε, ε, που θεωρεί πως μία παρέμβαση στο εθνικό δίκαιο είναι περιορισμένη προαιρετικό μέσο. Οπότε ε, τον ε, επεμβαίνουμε είναι οπωσδήποτε ε, πολύ πιο παρεμβατικό από το να προσφέρουμε ένα προαιρετικό μέσο. Και αυτοί που δεν το χρειάζονται, δεν το χρειάζονται, δεν είναι υποχρεωμένοι. Κάθε επιχείρηση μπορεί να πει, κοιτάξτε να δεν με ενδιαφέρει αυτό το προαιρετικό ευρωπαϊκό μέσο. Ε, δεν το χρησιμοποιεί κιόλα. Απλό είναι. Εάν όμως είχαμε ελάχιστη εναρμόνιση, θα έπρεπε Οπότε είναι σαφές πως είναι λιγότερο παρεμβατικός ο χαρακτήρας. Ή κάνω αυτό που, που ήξερα και δεν ασχολούμαι καθόλου με το νέο αυτό ευρωπαϊκό μέσο και τελείωσε. Για τη Ρώμη 1 τώρα υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις ε, προς όφελος των καταναλωτών. Παραδείγματος χάρη μπορούμε ως Γερμανοί καταναλωτές να πάμε στα γερμανικά δικαστήρια όταν ο αντίδικος, η επιχείρηση είναι, έχει ε, μια αντιπροσωπεία στη Γερμανία όπου να είναι. Ε, ε, αυτές οι εξαιρέσεις υπάρχουν ήδη και, και δικαιολογούνται νομίζω και είναι λογικές από την πλευρά προστασίας των καταναλωτών. Επί της ουσίας τώρα. Κι εγώ, εγώ συμφωνώ εδώ πέρα πρέπει λίγο να κάτσουμε πριν κάνουμε μεγάλες δηλώσεις και να τα διαβάσουμε. Αλλά ε, ένα είναι σημαντικό. Πρόκειται για μια πρόταση της Κομισιόν η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί αλλά έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από την θεωρία. Ε, εντάξει, είναι γνωστές ε, οι γνωμοδοτήσεις ειδικών, πανεπιστημίων, νομικών, αλλά εμείς Επιτροπή Προστασίας των Καταναλωτών. Θέμε να το κάνουμε φιλικό για τους καταναλωτές και στη διατύπωση ήδη δηλαδή. Εγώ συζητώντας και με τον κύριο Λένε είχα πρόθεση να μην είμαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι αλλά συνυπεύθυνοι. για να διαμορφωθεί πιο φιλικά προς τον καταναλωτή η αφετηρία. και βλέπετε πως ε, είναι λίγο δυσνόητο ορισμένα πράγματα, αλλά και εκεί πέρα με λίγες συμπληρώσεις ε, μπορούμε να ε, τα κάνουμε τα πράγματα πιο φιλικά προς τον καταναλωτή, να μην είναι ξέρα νομικά, να γίνει λίγο πιο κατανοητό. Γιατί οι νομικοί τα ξέρουν ήδη, εννοώ τους όρους και τους ορισμούς και όλα αυτά. Αυτό σε όλες τις χώρες. Η νομική γλώσσα δεν είναι η καθομιλουμένη viel äh, mitreden können, nicht Οπότε θα πρέπει νομίζω να μπορούμε να έχουμε και εμείς ένα λόγο σε ολόκληρο το κείμενο και την διατύπωσή του. Δεύτερον και ταυτόχρονα ερώτημα προς την Κομισιόν είναι εδώ ο κύριος Στάινμαϊρ, τον βλέπω. παρά το ότι υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των ε, καταναλωτών. Σε πολλές χώρες ε, εν μέρη υπάρχουν ε, κανόνες που διασφαλίζουν υψηλότερη προστασία. Εάν έχουμε την αρχή δικαίως πως όταν μια χώρα έχει υψηλότερο επίπεδο προστασίας τότε ισχύει το υψηλότερο επίπεδο, πρέπει να ε, γίνει εδώ πέρα φιλικότερο και για τις επιχειρήσεις. Το κείμενο αυτό. Τι θέλω να πω. Αν αντί για 27 καθεστώτα έχω ένα ευρωπαϊκό το δίκαιο το οποίο mm. επιλέγω πρέπει να καλύπτει όσο δυνατόν περισσότερα και όχι να προστίθεται και το εθνικό δίκαιο και να χρειάζομαι τελικά και το 28ο στο το ευρωπαϊκό και τα άλλα 27 που λέγαμε. Οπότε μπορούμε να έχουμε ένα παράρτημα το προτείνω αυτό προς την Κομισιόν και είναι μια παράκληση. Δηλαδή, να παρουσιάζονται οι υψηλότεροι ε, κανόνες προστασίας ε, στα κράτη-μέλη σε ένα παράρτημα. Ξέρω πως έχει ήδη γίνει προσπάθεια και είναι δύσκολο, αλλά τώρα νομίζω πως είμαστε πιο συγκεκριμένοι και μπορεί να γίνει η προσπάθεια. Έχουμε μια συνολική ωραία παρουσίαση ενός δικαίου συμβάσεων αγοράς και μπορούμε εδώ πέρα άρα έχοντας ένα επίπεδο να δούμε τις χώρες όπου είναι ε, υψηλότεροι οι κανόνες αλλιώς θα έχουμε δυσκολίες στην εφαρμογή δεν μπορεί και η μικρομεσαία επιχείρηση να λέει εγώ ε, επιλέγω το προαιρετικό δίκαιο αλλά τελικά στην πραγματικότητα δεν ξέρω ποιος θα ισχύσει. Δεν είναι λογική αυτή η κατάσταση. Και οπωσδήποτε θα πρέπει να ε, μιλήσουμε το, για το και να συζητήσουμε το εάν θεωρούμε λογικό ένα τέτοιο ε, παράρτημα. Ίσως μπορεί η Κομισιό να μας πει ορισμένα πράγματα ανεφικτό ένα τέτοιο παράρτημα έτσι ώστε πραγματικά να έχουμε ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό προαιρετικό σύστημα. Αυτά νομίζω φτάνουν, φτάνουν για σήμερα. Θα έχουμε και Υπάρχει λίγη ώρα ακόμα. Πρέπει, πρέπει να το συζητήσουμε λεπτομερώς. Ευχαριστώ πολύ. Yes, thank you very much. Uh, Πρόεδρος, σας ευχαριστώ και τους δύο. Βεβαίω θα πρέπει να συζητήσουμε για όποια τα θέματα, όμως ε, αυτά θα προκύψουν, ε, έχουν σχέση ακριβώ με αξιολογήσει. Ε, ευχαριστούμε και πάλι. Κύριε Μάντες, θα μιλήσετε στη θέση του κύριου Κρότσμαν. Ναι, ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε σχέση με το θέμα μας ότι τους αμέσως μήλυνες να συζητήσουμε την προστιθέμενη αξία. Όπως ανέφερε ο εισηγητής, πρόκειται για εκούσια ρυθμίση, Δεν εμπλέκονται και τα 27 κοινοβούλια όμως, παραμένει η δυνατότητα επιλογής. Σε περίπτωση λοιπόν που κάποιος δεν θέλει να προσχωρήσει αυτό το σχήμα. Έτσι μπορούμε να δούμε ε, το τι θα γίνει με συνεργασία. Πολλές φορές ε, δεν έχουμε μόνο με νομοθετικά εμπόδια, αλλά έχουμε το κόστος παράδοσης, γλωσσικό πρόβλημα. Τώρα, ε, σε σχέση με την επικοινωνία των επιχειρήσεων, Να πρέπει να δούμε γιατί δεν χρησιμοποιούν ε, ε επιχειρήσεις το σχήμα της απευθείας μεταξύ τους επικοινωνίας. Να δώσουμε μια, επεξεργα... μια ε, ευελιξία, να δούμε μήπως έτσι ε, θα μπορούμε να βάλουμε ακόμα ένα λιθαράκι στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα θεσπιστεί αυτό το νομοθέτημα με αυτή την εκούσια προσχώρηση, τότε αυτό θα είναι για όλους κάτι το ελκυστικό και θα μπορεί στην πράξη να χρησιμοποιηθεί. Έτσι μπορούμε να δούμε τις επιμέρους, ε, τους μεσορισμούς σε κάθε γλώσσα και στον περισσότερο καιρό ξεχνούμε τις ε, μικρομεσαίες. Υπάρχει με διάρκεια της τους. τώρα επιτέλους έχουμε μια θετική αντιμετώπιση. Έχουμε αυτόν τον ευρύτατο ορισμό. Και έτσι δίνεται η δυνατότητα εις όλες τις εταιρείες να προσχωρήσουν σε αυτό το σχήμα. Κατά αυτόν τον τρόπο δεν θα γίνεται διάκριση. Ε, βέβαια, μικρομεσαία επιχείρηση είναι και μια που μοιάζει σε όγκο με πολυεθνική, αλλά και ο μπακάρι τη γωνία. Το σχήμα προστασία επίση σημαντικό. Πάρα πολλέ είναι υποχρεώσει που τροβαρύνουν τι εταιρείε για να προσχωρήσουν στο νομοθέτημα. Ε, πολλέ επιχειρήσει δεν θα αποδέχονται δεν τους προσθέτει, δεν είναι την προστιμένη αξία, δεν θέλω να δεσμευτούν τόσο πολύ. Ότι επόμενες χρονισμού θα τα ξανασυζητήσουμε. Και αν τελικά ε, τέτοια ε, νομοθεσία ε, θεσπιστεί, θα, νομίζω ότι θα πετύχει. Και επίσης θα βελτιωθεί έτσι η εσωτερική αγορά. Αλλιώς θα είναι κρίμα όλη αυτή η δουλειά να πάει χαμένη. Άρα έτσι θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα από όσο είναι σήμερα. Ευχαριστώ. Πρώτα. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Είναι κρίμα το ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε την αξιολόγηση αντικτύπου με τον κύριο Στάτερμαϊρ. Εγώ εκτιμώ του ε, συνεισήγητε, αλλά η Κομισιόν εδώ πέρα δεν έχει κάνει μια εκτίμηση για το εάν χρειάζεται καν αυτή η πρόταση αν έχει εφαρμοστεί σωστά η οδηγία προστασία των καταναλωτών στα κρατη Τι θα γίνει όταν τεθεί ενισχύ η οδηγία. Και κάτι άλλο το οποίο δεν βλέπω εδώ πέρα καθόλου. Ξέρουμε πως το δίκαιο των πωλήσεων επηρεάζεται από αποφάσεις δικαστηρίων. Τι θα γίνει αν έχουμε αφενός αποφάσεις του ΔΕΚ και από την άλλη ε, νομολογία εθνικών δικαστηρίων. Τι θα γίνει Ποια είναι η σχέση μεταξύ των. Ε, πολλά ζητήματα λοιπόν άλυτα και δεν με ικανοποιεί η πρόταση της Κομισιόν. Και τέλος είναι εκπληκτικό το ε, πόσο μεγάλο είναι το μέτωπο της άρνησης και της απόρριψης από πολλά Και οι οργανώσει των καταναλωτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της βιομηχανίας είναι κατά. Και ε, τότε για ποιον κάνουμε αυτή την νομοθεσία άμα δεν τη θένε. Εγώ θα πω μόνο πως η ομάδα μας ε, και στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και εδώ πέρα ε, θα καταψηφίσει την οδηγία αυτή. Θα προσπαθήσουμε οπωσδήποτε να στηρίξουμε τους συγητές για περισσότερα δικαιώματα των καταναλωτών. Αλλά το αναφέρατε. Καλό αυτό το παράρτημα που λέτε για να ξέρουν τι γίνεται και στα κράτη-μέλη. Αλλά πούντο. Δεν μας το έδωσαν. Με ποια βάση νομοθετούμε λοιπόν εδώ πέρα. Ε, έχουμε κακή νομοθετική διαδικασία. Και, ε, κάτι τελευταίο, äh, είναι απολύτως απαραίτητο να ξεκαθαρίσουμε όταν προσπαθούμε για επιχειρήσεις και καταναλωτές να βελτιώσουμε τα πράγματα τι κάνουμε. Κανείς δεν θα χρησιμοποιήσει τελικά το δίκαιο αυτό εάν δεν υπάρξει μια βελτίωση. Στην δε εφατσέτ στην Frankfurt Allgemeine Zeitung μια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Κολονίας λέει κοιτάξτε δεν θα το διαλέξει κανείς αυτό καθώς οπότε και τι έγινε. Ε, ελπίζω να μην φτάσουμε εκεί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 για την πρόταση αυτή και την αξιολόγηση αντικτύπου ότι υπάρχουν σοβαρά μεθοδολογικά προβλήματα. Τα είχαμε πει αυτά και από την Πράσινη Βίβλο είχαμε ζητήσει μια αξιολόγηση αντικτύπου. Δεν τίποτα όμως δεν έγινε. Παραδείγματος χάρη Κομισιόν εδώ πέρα δεν λαμβάνει υπόψη το ότι πιθανώς κάποιος ο οποίος ε, ε, ο πελάτης ο διασυνοριακός και ο πολιτής ο διασυνοριακός ε, να δρά έτσι βάρος των εγχωρίων συναλλαγών. Γι' αυτό θεωρώ πως πρέπει οπωσδήποτε να γίνει συζήτηση. Επίσης τα κράτη-μέλη έχουν πολύ σοβαρές επιφυλάξεις όσον αφορά την ποιότητα αυτής της αξιολόγησης αντικτύπου και τα αποτελέσματά της και ζητήσαμε και εμείς στην Επιτροπή να λάβουμε σοβαρά και να εξετάσουμε σοβαρά την και οι οργανώσει των καταναλωτών εδώ πέρα θεωρούν πως η Κομισιόν δεν έχει δώσει τα κατάλληλα μέσα για να δικαιολογήσει την νομοθεσία αυτή και ζητάνε διαφορετικά μέτρα. Παραδείγματο χάρη μπορούμε να δούμε την πρόταση της BUC, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καταναλωτών για κάποια υποδείγματα συμβάσεων και ε, να υπάρχει η επιλογή. Άλλα σημαντικά επιχειρήματα όπως η οικονομική ανάπτυξη δεν τεκμηριώνονται εδώ πέρα από την Κομισιόν και πραγματικά αυτοί οι οποίοι θα υποφεληθούν καταναλωτές δηλαδή και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας λέει η Κομισιόν μα αυτοί είναι κατά ή να έχουμε λοιπόν ένα τόσο πολύπλοκο σύστημα, καλύτερα να κάνουμε μια ενημέρωση, θεωρώ εγώ. Και να τους πούμε ποιες είναι οι φυστάμενες διατάξεις και το τι σημαίνουν για τις διασυνοριακές πωλήσει ή το τι μπορεί να επιλέξει κανείς, τι κίνδυνοι υπάρχουν κτλ. Είμαι πεπισμένος και εδώ πέρα εκπροσωπώ και τον κύριο Φόξ πως χρειαζόμαστε την εσωτερική αγορά και η εναρμόνιση ε, θα χρησιμεύε και στην οικονομία μας. Δεν βλέπω όμως ε, το όφελος ε, στην εναρμόνιση εδώ πέρα των εθνικών συμβάσεων πολίσεων. Γιατί η επιλογή του ενδεδειγμένου δικαίου δεν είναι μόνο επιλογή του καταναλωτή αλλά και επιχειρήσεις. Θα πρέπει επομένω οι επιχειρήσει να έχουν περισσότερο περιθώριο, ούτω ώστε να μπορούν να αποφασίσουν. Να μπορούν να αποφασίσουν, λέγω. Διότι θα πρέπει τώρα να λάβουν υπόψη ότι υπάρχουν κάποιε χώρε με υψηλότερη προστασία του καταναλωτού. Α πούμε το Ηνωμένο Βασίλειο. Γι' αυτό και σα λέω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε όσον αφορά μια πρόταση ποιοτική, καλύτερη. Δεν νομίζω ότι με αυτή την πρόταση της Κομισιόν μπορούμε να πετύχουμε τους επιθυμητούς στόχους, διότι από την άλλη μεριά συνάδελφοι θέλουν εδώ να προστατεύσουμε καλύτερα, με πιο αποτελεσματική νομοθεσία τους καταναλωτές και να γίνει επίσης μια μελέτη επιπτώσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και έτσι να δούμε τα διαφορετικά σενάρια. Και ο κύριος Φόξ, επομένω ήθελε να απευθυνθεί εις τους εισηγητάς για να λάβουν υπόψη επίσης των των άλλων μέχρι ποιου σημείου μελέτη των επιπτώσεων είναι τεκμηριωμένη και τελικά να επιλεγεί η κατάλληλη, η καταλληλότερη, πρακτικότερη μέθοδος Επομένω, μπορώ παρά να πω στου συναδέλφου ότι θα πρέπει ψύχρεμα να κρίνουμε. Να λάβουμε υπόψη όλες τι απόψει και κυρίω απόψει των φορέων των καταναλωτών. Προσοχή. Να μην συμφωνήσουμε σε κάτι το οποίο αυξάνει τη γραφειοκρατία εις βάρος των επιχειρήσεων. να μην πάνε χαμένε τόσε διαπραγματεύσει όσον αφορά την οδηγία για του καταναλωτέ. Ο πρόεδρο. Κύριε Βαλτεσάρη, λίγο σκονοσμένοι, λάβανε εσεί το λόγο και κατόπιν εγώ θα συνοψίσω και να δούμε μετά με του σκιώδει ηγητά πώ θα προχωρήσουμε. Βαλτεσάρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομο. Νομίζω πω εντρέχουμε τον κίνδυνο να μπερδέψουμε τα πράγματα. Εδώ δεν πρόκειται για ένα νέο δικαίωμα των καταναλωτών. Πρόκειται για ένα μέσο επικαιροποίηση τη ενιαία αγορά που παρά την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, των ατόμων και των κεφαλαίων σε πολύ μεγάλο μέρος παραμένει νεκρό νεκρή. Ε, και στο ερώτημα γιατί δεν λειτουργεί, δεν έχει ενεργοποιηθεί πλήρωση η νέα αγορά, ε, πολύ συχνά έχουμε ως απάντηση την έλλειψη ενός νομικού πλαισίου που να εγγυάται με, με όμορφο τρόπο τις συμβάσεις εκτός από τη γλώσσα, τις διαφορετικές ε, συνήθειες, ηθικές κτλ. Ναι. Άρα λοιπόν, εδώ δεν έχουμε σχέση μεταξύ επιχείρηση και καταναλωτή, άρα επιχείρησης και επιχείρηση Ιταλική και Σουλβακικής, α πούμε. Διαφορετικές παραδόσεις, διαφορετικά νομικά συστήματα. Και επειδή δεν μπορούμε να εναρμονίσουμε 27 ε, διαφορετικά εμπορικά δίκαια, ε, μόνο, μόνη λύση, αν δεν θέλουμε να υιοθετήσουμε τα μέσα του διεθνούς δικαίου, τα, τα εργαλεία του διεθνούς δικαίου, να βρούμε ένα προαιρετικό δίκαιο, το οποίο δεν είναι... Δεν ακυρώνει ε, δεν είναι δηλαδή μια ανακοίνωση κάποιων ε, προθέσεων. Μιλάμε για 150 άρθρα. Μιλάμε για το θέμα το ποιο είναι υπεύθυνο που δεν ανταποκρίθηκε στην κάποια υποχρέωση, το δικαίωμα άρνηση του προϊόντο, ευθύνη του φόρε... ευθύνη του αποστολέα κτλ, κτλ. Το δίκαιο των πωλήσεων σε όλε τι πτυχέ του. Γιατί, ε, γιατί δύο επιχειρήσει ε, ή ένα επιχειρηματία και ένα καταναλωτή να μπορούν να επιλέξουν ποιο είναι το δίκαιο που διέπει τη σχέση του με συγκεκριμένο και σαφή τρόπο με υποχρεώσει και δικαιώματα πολύ καλά καθορισμένα. Το 33% των αγορών γίνεται πλέον μέσω του ίντερνετ μέσα στα κρατημέλη. Όταν όμως πρέπει να γίνουν αγορές διασυνοριακά, πέφτουμε στο 7%. Γιατί, Γιατί ο καταναλωτής δεν έχει εμπιστοσύνη. Εγώ αγοράζω 100 μπουκάλια κρασί, ας πούμε, από έναν Ιταλό έμπορο και άμα δεν μου τα στείλει ποιος πληρώνει. Και αν πληρώσω, πληρώσω και δεν μου φτάσει το με τα κάνω. Α, μεγάλα ερωτήματα και εμπόδια για μια πλήρη ανάπτυξη της εσωτερικής ενιαίας αγοράς. Αυτό το μέσο λοιπόν είναι το μόνο ή μάλλον είναι ένα από τα μέσα που μας επιτρέπει να ευνοήσουμε τις εμπορικές αλλαγές δια, ε, κρατικά. Και η προστασία του καταναλωτή είναι πολύ ψηλή. Ίσως σε ορισμένε χώρε να προστατεύεται ακόμη περισσότερο ο καταναλωτή. Αλλά σίγουρα υπάρχει μια βάση επί τη οποία ε, να συμφωνήσουμε. Ήδη είναι εξαιρετικά συγκεκριμένη και ευρεία αυτή η βάση. Και η προστασία του καταναλωτή προστατεύει μάλλον τον καταναλωτή σε όλες τις περιπτώσεις. Γι' αυτό και θα ήθελα και να αξιολογήσουμε την υπόλοιπη συζήτηση. Δεν είναι ακόμα ένα δικαίωμα του καταναλωτή. Είναι ένα μέσο που επιτρέπει στον καταναλωτή να αγοράζει και έξω από τη χώρα του. Γιατί Διαφορετικά οι επιχειρήσει γίνονται θύματα τη παγκοσμιοποίηση και δεν τη χρησιμοποιούν όμω δεν εκμεταλλεύονται τη, δυνατότητα διεθνοποίηση που γίνεται μέσω τη δυνατότητα πώληση εκτό τη χώρα και εκτό τη περιοχή. Εάν δεν εγγυηθούμε τέτοιου είδου δικαίωμα, δεν είναι δυνατόν να έχουμε μέσα που να βοηθούν αυτέ τι ανταλλαγέ και να καθιστούν αποτελεσματική την ενιαία αγορά. Γι' αυτό λοιπόν με κάθε δυνατή βελτίωση πιστεύω πως είναι μια λύση βεβαίως που μπορεί να βελτιωθεί, επιδέχεται βελτίωση, αλλά μια κεντρική λύση με την οποία θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια από νομοθετικής άποψης, εμπόδια που ακόμα δυσχεραίνουν την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς. Πολύ ζωντανή θα είναι η συζήτηση για αυτό το θέμα. Και ο κ. Βαλτασάρα έχει δίκιο ότι σίγουρα αυτό προτείνεται ω ένα εργαλείο για τη βελτίωση των δυσυνοριακών πωλήσεων, για την αύξηση των δυσυνοριακών πωλήσεων. Αλλά υπάρχουν και άλλα μέσα που το κάνουν το αυτό και φυσικά η οδηγία για τα δικαιώματα του καταναλωτή, αν εφαρμοστεί σωστά, είναι σημαντικό βήμα προ κάτι τέτοιο. Τώρα μας τελείωσε ο χρόνος. Δεν θα σας ακούσουμε τον κύριο, τον αρμόδιο την Επιτροπή, γιατί αλλά ξέρω πως μας άκουσε με ενδιαφέρον. Προσπαθήσω να συναψίσω και να προτείνω πώς να προχωρήσουμε. Κανονικά θα αρχίσουμε τη συζήτηση για μια νέα πρόταση μέσω της αξιολόγησης ε, αντικτύπου της Κομισιόν που δεν μπόρεσαμε να το κάνουμε γιατί χρειαζόμαστε ακόμα μια ώρα ή λίγο ακόμα για να το κάνουμε αυτό. Και επίσης πιστεύω ότι οι συγητές και οι σκιώδεις θα πρέπει να με ποια μορφή θα γίνουν όλα αυτά. Ήδη ακούσατε διάφορους συναδέλφους που έθιξαν το ερώτημα, που ήδη έχουν αλλά διαβάσει την εκτίμηση αντικτύπου. Θα είναι μακρά η συνεδρία λοιπόν. Ίσως να θέλετε κύριοι συγητές να σκεφτείτε μήπως ε, θέλετε να ρωτήσετε από τη μονάδα που έχουμε τη μονάδα αξιολόγησης επιπτώσεων να μελετήσει την έκθεση της Επιτροπής και να κάνει και παρατηρήσεις. Πάμπλο, λίγο πιο σιγά σε παρακαλώ. Μπορείς να μιλάς λίγο πιο σιγά γιατί σε ακούω. Μπορείς να, ή να, αλλιώς να περάσεις έξω σε παρακαλώ. I think that, uh, if I could ask the rapporteurs to get together with the shadow rapporteurs, I think it's been an important... Νομίζω λοιπόν πως ήταν μια σημαντική πρώτη ανταλλαγή απόψεων γιατί αποδεικνύει τις διαφορές προοπτικής και σαφώς θα πρέπει αυτές να τις λάβουμε υπόψη. Πρότασή μου είναι λοιπόν να έχουμε μια συνεδρία ολόκληρη για την ε, αξιολόγηση αντικτύπου και να το στέλνουμε να τη μελετήσουμε εις βάθος Αυτή είναι λοιπόν η πρότασή μου. Και θα είναι λίγο διαφορετικό το project λόγω της συνεργασίας των δύο εισηγητών. Νομίζω πως θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια καλή συμφωνία με την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων που νομίζω ήδη το είδατε αυτό ως βάση. Καταλαβαίνω τα όσα είπε η κυρία Γκέμπχαρτ αλλά αν η Κομισιόν, μάλλον η Επιτροπή μας επιθυμεί να προτείνει διαφορετικές λύσεις, μπορεί να το κάνει. Και θα βρούμε τρόπους όλα αυτά να τα εντάξουμε στη δομή της πρότασής μας. Θα είναι σημαντικό αυτό. Περισσότερο για διαδικαστικά θέματα ήθελα να μιλήσω και όχι για την ουσία. Δεν ξέρω αν θέλει ο κ. Μάγερ, η κυρία Γκέπχερ θέλουν να κάνουν κάποιες σύντομες παρατηρήσεις. Πέντε λεφτά είχαμε, σχεδόν τα έφαγα εγώ. Μήπω όμω θέλετε παρόλα αυτά να κάνετε κάποια τελευταία παρατήρηση, ο κύριος, ο Μάγερ. Σύντομα. Πρέπει να λειτουργήσει καλύτερα η ιστορική αγορά. Η Επιτροπή Νομικής Νομικών Υποθέσεων έχει άλλη δουλειά. Δηλαδή έχουμε πολλούς νόμους. Διάφορα πράγματα. Ευρωπαϊκά εντάλματα. Διάφορα πράγματα. Αλλά δεν υπάρχει ουσιαστική ευρωπαϊκή νομοθεσία για το τι συμβαίνει, πότε πραγματικά συνάπτεται μία σύμβαση, ποιες οι συνέπειες αυτής, τι γίνεται όταν δεν εφαρμόζεται. Αν δηλαδή αν τα παίρνουμε σοβαρά και λέμε ότι έχουμε εσωτερική αγορά, ο καθένας λέει και αγοράζει όπου θέλει, όπως θέλει, ε, πρέπει αυτά τα πράγματα να λειτουργούν. Αυτό πρέπει να σκεφτούμε και να εγκρίνουμε. Τα υπόλοιπα τα συζητάμε. Ε, τα βασικά στα οποία συμφωνούμε όλοι. Ε, χρειαζόμαστε βασική προσέγγιση τι θα γίνεται σε μια ιστορική αγορά για να μπορεί να λειτουργεί και να πουλάει και να αγοράζει ο καθένας. Επίσης, δεν μπορώ να ακούω πράγματα του στυλ ή ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι κατά. Κοιτάξτε, το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο στη Γερμανία είναι υπέρ. Ποιο ρωτήσατε εσείς και λέτε το απορρίπτουν όλοι. Το, το ενέκριναν στο, στο εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο στο Βερολίνο. Πριν από τρει εβδομάδε που ήρθα σε επαφή μαζί του. Και τέλος... Wenn man das optionale Recht Αν επιλέξουμε κάτι το προαιρετικό, να ισχύει πάντα παρόλα αυτά το ε, υψηλότερο επίπεδο προστασίας. Να μην υπάρχει ο φόβος ότι θα μειωθούν ε, τα δικαιώματα των καταναλωτών. Όχι. Όχι. Αναφέρεται. Σε περίπτωση εμφωλίας ισχύει το υψηλότερο επίπεδο προστασίας. Τέλος. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε ένα παράρτημα για να μπορεί κανείς να διαβάσει τα υψηλότερα επίπεδα προστασίας που δεν καταργούνται. Τέλος αν θα γίνει τώρα αυτή η συζήτηση, θα γίνει άλλη ώρα, δεν, λέω άλλα. Βεβαίω ε, τώρα μπήκε στον πειρασμό και η κυρία Γκέμπχαρτ να πει την τελευταία λέξη. Ε, δεν θα τα αφήσω αυτό να περάσει έτσι αυτό το οποίο ακούστηκε. Εμένα μου πάνε άλλα πράγματα από το επιμελητήριο. Ναι. Δεν ξέρω με ποιον μιλήσατε εσείς. Άλλοι μιλήσαμε με μένα, άλλοι μιλήσαμε με τον Χάνς Πέτερ. Ενδιαφέρον. Αλλά πρέπει να συζητήσουμε με ποια μέσα θέλουμε να επιτύχουμε να λειτουργεί η κοινή ιστορική αγορά με υψηλό ποιοτικό επίπεδο. Αυτό είναι το θέμα μας. Και μπορεί να γίνει με άλλους τρόπους που δεν πρέπει να παραμελήσουμε. Όταν ακούω δηλαδή, ε όχι, όταν ακούω ε, επιχειρήματα του στυλ ε, θα ισχύσει παρόλα αυτά το υψηλότερο επίπεδο προστασίας, ε, τότε δεν το χρειαζόμαστε καθόλου αυτό το μέσο εδώ πέρα. Δεν έχει προσθέμενη αξία. Τώρα, τώρα, τώρα δεν θα ξεκινήσει η συζήτηση μεταξύ των εισηγητών. Αυτό το οποίο έδειξε η συζήτηση είναι πως δεν υπάρχει συνένεση ούτε εδώ μέσα, ούτε στο Συμβούλιο, ούτε σε οργανώσεις ε, καταναλωτών και βιομηχανίας. δουλειά μας λοιπόν είναι να εργαστούμε συστηματικά όπως κάνουμε στην Επιτροπή μας για να ε, έχουμε ένα λογικό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν. Ευχαριστώ την Κομισιόν και βεβαίως ε, αναμένω τα επόμενα βήματα από τους εισηγητές. Η επόμενη συνεδρίαση είναι 25 και 26 Απριλίου το πρωί. Ευχαριστώ. Some extra time and I look forward to seeing you in Strasbourg next week.